Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Να αρχίσουμε αμέσω τη συνεδρίασή μας για σήμερα το απόγευμα. Πρόκειται για τη δημόσια ακρόαση με θέμα η κρίση στη Συρία και ο ρόλος των διεθνών και περιφερειακών παραγόντων. Επιπτώσεις στην ασφάλεια για την Ευρώπη. Είναι τιμή για μένα που μπορώ να καλωσορίσω εδώ τους εξέχοντες προσκεκλημένους μας, την κυρία Βιζινή, Διευθύντρια Πολιτικής Ασφάλειας και Πρόληψης Συγκρούσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ο δεύτερος είναι ο Εμίλ Χοκεγέμα, που είναι Senior Fellow του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών ε, Μελετών για τη Μέση Ανατολή, τον κύριο Μάικλ Μπεναμού, ο οποίος είναι ερευνητής στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών Βίλφριντ Μάρτενς. Η κυρία Ζενή μας έρχεται κατευθείαν από το αεροπλάνο και ο κύριος Χόκεγεμ από ό,τι έμαθα βιάζεται γιατί και αυτός έχει να πάρει ένα αεροπλάνο. Οπότε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Χοκαγιάμ. Μετά στην κυρία Ζενή και τέλος στον κύριο Μπεναμού. Εντάξει, παρακαλώ. Κύριε Χοκαγιάμ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Είναι τιμή για μένα και ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Πρέπει να φύγω λίγο νωρίτερα γιατί πράγματι πρέπει να πάρω αεροπλάνο να επιστρέψω στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να ξαναβρεθώ στην περιοχή για να ξαναβρεθώ μέσα στα πράγματα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας παρουσιάσω κάποια σημεία για να υπάρχει μετά χρόνος για συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, υποτιμήσαμε πάρα πολύ το μέγεθος και τη σημασία της Συριακής κρίσης και τις ανθρωπιστικές της επιπτώσεις και αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα όσα έγιναν εκεί δεν ήταν απλώς προβλεπόμενα, είχαν ήδη προβλεφθεί. Για πολλούς και κατανοητούς λόγους. Υπήρχε κούραση από το Ιράκ, από την Αραβική Άνοιξη είχαμε καταλήξει στο ότι ο αραβικός κόσμος είχε πέσει στην απελπισία, δεν υπήρχε ελπίδα από εκεί. Δεν καταλάβαμε λοιπόν καλά ούτε την κρίση ούτε τις επιπτώσεις της. Και είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα θα έλεγα αντίδρασης ε, με σύγχυση και εφαρμογή πολιτικής μέσα σε σύγχυση. Τώρα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε καλύτερα την δυναμική της σύγκρουσης αυτής. Ο πόλεμος στη Συρία που ξεκίνησε σαν επανάσταση και κατέληξε σε εμφύλιο πόλεμο κατέστρεψε τη Συρία. Τα γνωρίζετε τα νούμερα. 5 με 6 εκατομμύρια είναι οι πρόσφυγες, 7-8 μετατοπισμένοι εκατομμύρια. Η κατάσταση επί τόπου είναι τραγική με τις μαζικές μετακινήσεις. Επίσης ο πόλεμος στη Συρία άλλαξε και τη ζωή των γειτόνων της διότι υπάρχουν επιπτώσεις διάφορες όπως για παράδειγμα τα συγκρόμενα ε, μέρη φτάνουν μέχρι το Ισραήλ δημογραφικά αλλάζει η κατάσταση στην περιοχή, οι κοινωνίες, τα σύνορα ίσως, το πώς οι χώρες, τα κράτη αντιλαμβάνονται τη δικιά τους ασφάλεια και τη θέση τους στην περιοχή. Είναι λοιπόν ένας πόλεμος, μια σύγκρουση που έχει επηρεάσει και την Ευρώπη και αυτό θα το συζητήσετε περισσότερο με τον συνάδελφο. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι ποτέ δεν ήταν μια σύγκρουση που μπορούσαμε να καθορίσουμε συγκεκριμένα. Πριν από χρόνια ο κόσμος θεωρούσε ότι τη σύγκρουση στη Συρία μπορούσαμε να την περιορίσουμε. Ίσως επειδή είχαμε δει τι έγινε στο Ιράκ, επειδή υπήρχε η Αμερικανική παρέμβαση στο Ιράκ το Ιράκ ε, το βλέπαμε σαν τον μεγάλο εφιάλτη. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι κάτι θα πάει χειρότερα από ότι πήγαν τα πράγματα στο Ιράκ. Ε, λοιπόν, πήγαν στη Συρία. Χωρί να σημαίνει ότι μία περίπτωση είναι καλύτερη ή χειρότερη, δεν είναι αυτό που θέλω να πω για τι συγκρούσει, Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι επιπτώσει είναι μεγαλύτερε. Συνεπώ χρειάζεται στρατηγική σαφήνεια για το τι συμβαίνει εκεί. Και μια που βρίσκομαι στι Βρυξέλλε και δεδομένα το γεγονότο του τελευταίου μήνε και χτες και σήμερα μάλιστα πιο συγκεκριμένα, πρέπει να σας πω ότι όταν μιλάμε για τη Συρία επικεντρωνόμαστε πολύ στους πρόσφυγες και στο λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Είναι απόλυτα κατανοητό και δικαιολογείται σε έναν βαθμό, αλλά από πλευρά Μέση Ανατολή, από πλευρά τη περιοχή εκεί δηλαδή, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μα ότι ο Ασάτ και το καθεστώ του αποτελεί την κύρια αιτία θανάτων και μετατόπισης πληθυσμών. Και με τον Ασάτ τα έχει βάλει κυρίως η Δύση, τον βαρδίζοντας και τα λοιπά. Όχι τόσο το Ισλαμικό κράτος. Αντίδραση εκτός μικροφώνου από την αίθουσα. Εγώ δίνω το λόγο, λέει η Πρόεδρος. Δεν σας έχω δώσει το λόγο, λοιπόν. Συνεχίζει ο Να το τονίσω. Στον Ασάντ οφείλονται οι περισσότεροι θάνατοι στην περιοχή και τα προβλήματα. Οι πρόσφυγες εξάλλου δεν πηγαίνουν στο Καλυφάτο, πράγμα το οποίο τι δείχνει. Δείχνει ότι το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος δεν είναι ελκυστικό για τον κόσμο στην περιοχή. Αυτό που εννοώ είναι ότι η ανθρωπιστική κρίση δεν είναι η ατυχής συνέπεια της σύγκρουσης είναι μια στρατηγική του καθεστώτος του Ασάντ με πολλές πτυχές. Το καθεστώς του Ασάντ λοιπόν υιοθέτησε τη στρατηγική κλιμάκωσης από το 2011 και μετά. Και ξέρετε είναι σαφές το μήνυμα της καταστολής, της λιμάκωσης αρχίζεται με ε, μικρά προβλήματα, κάποιες μικρές μάχες, μετά σιγά σιγά βάζετε και τα βαλιστικά, μετά και ε, πυρηνικά όπλα ή ξέρω εγώ μαζικής καταστροφής κτλ. Και άρχισε να το κάνει. Και έτσι έγινε πιο κατάσταση ακόμα. Το δεύτερο σκέλος της στρατηγικής αυτής του Ασάντ είναι να κυκλοφορεί η πληροφορία και η άποψη ότι εδώ πέρα πρόκειται από τη μια μεριά ο Ασάτ και από την άλλη μεριά οι ακραίοι. Ο κόσμος το πίστεψε συχνά, αγνώντας την πραγματικότητα. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας της Συρίας δεν στηρίζει τον Ασάντ ούτε τους ακραίους και οι εχθροπραξίες τις τελευταίες εβδομάδες ακριβώς αυτό έδειξαν. Έδειξαν την αντοχή ενός κέντρου μετριοπαθούς της Συριανής ε, κοινωνίας που δεν είναι ούτε με τους μεν ούτε με τους δε. Τα βάζουν και με το Ισλαμικό κράτος και με τον Αμπάσαρούσα. Είναι λοιπόν μια επίτηδες στρατηγική αυτή. Το καθεστώς του Ασάντ δεν προσπαθεί να κερδίσει και πάλι τις καρδιές και τα μυαλά των ε, πιστών πολιτών. Προσπαθεί είτε να τους σκοτώσει είτε να τους διώξει από τη χώρα. Και το βάρος, την ευθύνη την αποδίδει στους αντιπάλους του ή στους ε, δυτικούς. Και έτσι παραλύει η δυνατότητα για αποφάσεις. δεν αντιμετωπίζεται η ανθρωπιστική κρίση. Και αυτό είναι πολύ βασικό εδώ που θέλω να σας πω, ότι η ανθρωπιστική κρίση δεν είναι το ατυχές αποτέλεσμα της σύγκρουσης. Όχι, είναι η στρατηγική του Ασάντ, που το πολιτικό κεφάλαιο, του πόρους, το χρόνο του δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει, γιατί δεν νομίζω και ότι μπορεί, για να κερδίσει πίσω τον κόσμο. Όχι, γι' αυτό και τους διώχνει. Ας κοιτάξουμε λίγο πιο συγκεκριμένα το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Η ηρωνία και τραγωδία είναι ότι το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος είναι εχθρός των πάντων. Όλοι θεωρούν ότι το ISIS είναι ο εχθρός τους. Και μόνο το Ηνωμένο Πολιτειών είναι προτεραιότητα και όσων βρίσκονται βέβαια επί τόπου και των Ευρωπαίων που ασχολούνται με αυτό. Οπότε αν είσαστε με τον Ασάτ, τα βάζετε με τους αντιστασιακούς. Βλέπετε τον Ασάντ πιο πολύ από ότι το ISIS τελικά. Τον βλέπετε σαν μεγαλύτερο αντίπολο. Αν είσαστε στην Τουρκία μπορείτε να θεωρείτε ότι η μεγαλύτερη απειλή είναι η επιθυμία των Κούρδων. Και άρα θεωρείστε ότι συνεργάζεστε με το ISIS. Ή μπορεί αν το δείτε από άλλη πλευρά, ε, οι Αμερικανοί να βάζουν προτεραιότητα αλλού, στην Ιεμένη, δεν ξέρω εγώ αλλού. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένα ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Και αυτό εξηγεί σε ένα βαθμό γιατί αυτό το τέρας των τζιχατιστών παραμένει. Δεν ενισχύεται, δεν αποδυναμώνεται, τροποποιείται. Και δεν πρόκειται να σταματήσει με τη συνηθισμένη μας μέτρηση του κατά πόσο ανεβαίνει η δύναμή του ή κατεβαίνει. Όχι. Παραμένει μεταμορφόμενο. Ας θυμηθούμε το Ιράκ στις αρχές καταπολέμησης του ISIS. Η στρατηγική στο Ιράκ ήταν τέτοια που η γεωγραφία και η δημογραφία δεν βοηθούσε το ISIS γιατί μπορεί να άρεσε στο 20% το πολύ του πληθυσμού, οι οποίοι όμως βρισκόντουσαν από τη Βαγδάτη στην ε, Μουσούλη και από την ε, Βαγδάτη ανατολικά ε, στα μέρη που δεν είναι τα πιο καλά και τα πιο πλούσια του Ιράκ. Δεν λέω ότι το 90% του πληθυσμού θα τα βάζε με το ISIS, αλλά πάση περιπτώσει δεν ήταν υπέρ. Ενώ περίπου 70% του πληθυσμού βρίσκεται αλλού στη Συρία. Βέβαια τα καλά νέα όταν μιλάμε για το Ισλαμικό κράτος στη Συρία είναι ότι υπάρχουν εναλλακτικέ. Οι πρόσφυγες αυτοί οι οποίοι φεύγουν από τη Συρία δεν πηγαίνουν στο Καλυφάτο γιατί το Καλυφάτο έχει ελάχιστα πράγματα να προσφέρει και αυτή είναι μια βασική αποτυχία του Ισλαμικού κράτους. Στο Ιράκ το καλό είναι ότι το Ισλαμικό κράτος δεν μπορεί να πολεμήσει όπως στη Συρία. Κάτι άλλο είναι ότι η Συριακή σύγκρουση ε, είναι και σε ολόκληρη την περιοχή, αλλά έχει πάρει και ένα διεθνή χαρακτήρα και τι εννοώ αυτό, ότι η Ιρανοί, η Σαουδική Αραβία είναι παράγοντες στη σύγκρουση αυτή. Καταστροφικοί παράγοντες βέβαια. Έτσι έχει υπάρξει πόλωση στην κοινωνία και η συμφιλίωση έχει καταστεί πάρα πολύ δύσκολη. Είναι και μια σύγκρουση επίσης που διεθνοποιήθηκε ιδιαίτερα από το Σεπτέμβριο που παρενέβησαν οι Ρώσοι. Γιατί αυτή η ρωσική παρέμβαση ήταν και στη διπλωματία αλλά και στις ε, μάχες. Ευνοεί τον Ασάντ βραχυπρόθεσμα και η Ρωσία φάνηκε ότι ε, συμπεριφέρθηκε με τρόπο που εξέπληξε ακόμα και τον Αμερικανό πρόεδρο. Και θα δούμε πόσο θα συνεχιστεί. Τα αποτελέσματα υπέρ όμως της Ρωσίας ήταν πολλά γεωπολιτικά, αλλά και για την ε, Συρία, γιατί επιβιώνει ο Ασάντ, βρίσκεται στο κέντρο της διπλωματίας και νομίζω μάλιστα ότι όσον αφορά τη Ρωσία αυτό που θέλουν είναι μια παγωμένη σύγκρουση και όχι ένα διακανονισμό. Και ίσως το καταφέρουν. Είναι μια διεθνή σύγκρουση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δευτερεύοντα ρόλο. Παίρνει τους πρόσφυγες, ξοδεύει δισεκατομμύρια. Αλλά δεν αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη σύγκρουση που βρίσκεται στα σύνορά της και που επηρεάζει την δικιά της συνοχή και ασφάλεια. Κάποιες χώρες είναι πολύ αυστηρές απέναντι στον ε, Ασάντ, άλλοι προτιμάνε τον Ασάντ από ότι το Ισλαμικό κράτος, αλλά αυτή είναι μια επιλογή δεν είναι πραγματική επιλογή. Η διπλωματία τώρα σήμερα, για να δούμε. Εγώ δεν είμαι κοινικός, είμαι σκεπτικιστής. Οπότε περιμένω να δω στη Γενέβη τι θα πετύχουν οι διαπραγματευτές. Όμως το ζήτημα είναι να καταλάβουμε ότι η πρόοδος ή αυτό που λέμε πρόοδος στην Γενέβη το 2544 ψήφισμα κατέστη δυνατό εξαιτία δύο παραγόντων. Πρώτον, επειδή οι Ηνωμένε Πολιτείε περιόρισαν τους πολιτικούς τους στόχους και αποφάσισαν απλώς να μην στηρίξουν τις πλευρές που είχαν πει ότι θα στηρίξουν για ένα διάστημα τουλάχιστον και ζήτησαν από τους συμμάχους τους να προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση. Εγώ νομίζω ότι είναι λάθος, αλλά πάση περιπτώσει απλώς το περιγράφω τώρα. Το άλλο, το οποίο βοήθησε τη διπλωματία να προχωρήσει, είναι η Ρωσία. Είναι η πολιτική και στρατιωτική παρέμβαση της Ρωσίας που διαμόρφωσε τα πεδία της μάχης. Η Ρωσία σήμερα εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη δύναμη Ακόμα και η απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας που ανακοινώθηκε αποτελεί μοχλό στα χέρια της Ρωσίας. Ο πρόεδρος Πούτιν που δεν τον περιέγραφαν πολύ κολακευτικά οι άνθρωποι για ένα διάστημα, αλλάζει. Ακόμα και αν πολλοί εδώ στην αίθουσα δεν συμφωνούν. Η κατάσταση λοιπόν είναι πολύ περίπλοκη. Η Ρωσία έχει διασφαλίσει την παρουσία του ασατ και διατηρεί τη δυνατότητα να επιστρέψει για να τον στηρίξει αν χρειαστεί. Συγχρόνως οι Ηνωμένε Πολιτείε κρατάει την Ανατολική Συρία. Εκεί δηλαδή που βρίσκεται το Ισλαμικό κράτος, το πιο δύσκολο κομμάτι. Ο πρόεδρος Πούτιν είπε ότι δεν πήγε στη Συρία για να πολεμήσει το Ισλαμικό κράτος. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Ποτέ δεν πήγε στη Συρία για να αποδυναμώσει τον τζιχαντισμό. Πήγε για να σώσει τον Ασάντ. Και όσον αφορά την κατάπαυση πυρός, είναι καλό ανθρωπιστικά. Αλλά μην υπερβάλλουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν σήμερα. Ο Ασάντ δεν επιτρέπει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε διάφορες περιοχές που βρίσκονται ακόμα σε Πολιορκία. Βέβαια, μα ικανοποιεί το ότι περισσότερο κόσμο έχει πρόσβαση σε τρόφιμα και σε φάρμακα, αλλά έτσι όπω χρησιμοποιείται αυτή η αμφισημία από τον Ασάντ, δεν έχουν σταματήσει εντελώ ούτε οι μάχε. Αυτό που είδαμε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες είναι ότι οι εχθροπαξίες, οι εχθροπραξίες, οι τους βοήθησαν να προχωρήσουν ο Πούτιν και ο Ασάντ σε κάποιες περιοχές. Συνεπώς, υπάρχει λόγος για ελπίδα, αλλά υπάρχουν και παρενέργειες με την κατάπαυση αυτή πυρός. Συνεπώς, το στοιχείο κλειδί είναι η μετάβαση, η τύχη του Ασάντ να εξακολουθεί να συζητιέται. Αλλιώς, καταλήγουμε με μια απαγωμένη σύγκρουση που βέβαια σήμερα φαίνεται κάτι θετικό σε σύγκριση με την ανθρωπιστική κρίση αλλά θα οδηγήσει σε νέες συγκρούσεις και σε επιπτώσεις όχι μόνο στην άμεση γειτονία της Συρίας αλλά ακόμα και εδώ στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να παρακαλέσω την κυρία Ζένη να κάνει την παρέμβασή της. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε εδώ πέρα αλλά και που οργανώσατε τη σημερινή συζήτηση. Η Συρία αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές τραγωδίες που έχουμε δει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όσον αφορά τον αριθμό των εκτοπισμένων. 6,5 εκατομμύρια ε, ανθρώπων από τη Συρία έχουν εκτοπιστεί και Υπάρχει μεγάλος αριθμός αυτών που δεν έχουν πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε το κρίσιμο αυτό θέμα. Θα ήθελα κατά κάποιο τρόπο να συμπληρώσω την παρουσίαση που, ακούσουμε, που ακούσαμε, να επικεντρωθώ περισσότερο στον τίτλο της συζήτησης που είναι ο αντίκτυπος στην ευρωπαϊκή ασφάλεια που είναι ε, θέμα που με αφορά και μένα πιο πολύ στην ε, ιδιότητά μου ως ε, Διευθύντρια της Πολιτικής Ασφαλείας. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω τη δική μου εικόνα για την πολύπλοκη αυτή κρίση και να σας πω τι κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε. Όπως ακούστηκε, το κεντρικό θέμα είναι η πολιτική διαδικασία. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Πολλοί κόσμος υποτιμάει την πολυπλοκότητα του θέματος και τη σημασία της προόδου στο πολιτικό σκηνικό, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση από μια πολιτική επίλυση του προβλήματος με επικεφαλής τους ίδιους τους σύρους. Φυσικά, αναφέρθηκε ότι μια από τις πιο σημαντικές διαστάσεις της σύγκρουσης στη Συρία όταν κοιτάμε το αντίκτυπο στην Ευρώπη είναι ο ρόλος του Ντάες στο σύνολο της εικόνας. Η Ντάες είναι δημοφιλής σε όλο τον κόσμο έχει χρησιμοποιήσει με πολύ ικανό τρόπο τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Έχει κάνει πολύ καλή προπαγάνδα, έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο μια πολύ καλή μάρκα, ένα πολύ καλό όνομα ε, και έχει κερδίσει έδαφος από τη Σομαλία στον Μπαγκλαντές μέχρι και τις Φιλιππίνες. Τούτου λεχθέντος δεν πρέπει να υποτιμούμε το γεγονός ότι και η Αλκάιδα παραμένει απειλή. Είναι λοιπόν ε, πολύπλοκη η εικόνα όσον αφορά την ε, ευρωπαϊκή ασφάλεια από πλευρά της τρομοκρατίας. Τούτου λεχθέντος θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αν κοιτάξουμε τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη ε, πραγματοποιήθηκαν κυρίως από ανθρώπους που έχουν γεννηθεί εδώ και από τρομοκρατικούς πυρήνες εντός της Ευρώπης. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι σε πολλές άλλες συζητήσεις όταν εξετάζουμε την τρομοκρατική απειλή από τη Ρωσία υπάρχει τάση και κίνδυνος να εξισώνουμε την μεταναστευτική κρίση που ήδη περιγράφει και δεν θα επαναλάβω όσα ήδη υπόθηκαν. Ε, υπάρχει λοιπόν κίνδυνος να συγχαίουμε αυτό με την ε, εικόνα της τρομοκρατίας εντός της Ευρώπης. Γιατί μια τρομοκρατική ομάδα να θέλει να χρησιμοποιήσει τις μεταναστευτικές οδούς στη στιγμή που είναι ε, δρόμοι μη ασφαλείς, δεν μπορούν να φέρουν μαζί τους εξοπλισμό και εάν δούμε τις επιθέσεις στο Παρίσι, αυτές οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από ανθρώπους εντός της Ευρώπης. πώς θα προχωρήσουμε. Κρίσιμο είναι να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες του προβλήματος. Ποιοι είναι οι παράγοντες που προκαλούν ανασφάλεια στην Ευρώπη. Χρειάζεται λοιπόν πολιτική επίλυση της σύγκρουσης εντός της Συρίας καθώς και στην Λιβύη και στα Παλαιστινιακά εδάφη. Βλέπετε είναι θέματα που ε, ανακύπτουν συνεχώς ε, στο θεματολόγιο. Όλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος της ευρύτερης προσέγγισής μας ε, και της συνεργασίας μας με τις χώρες της περιοχής, τις συμφωνίες σύνδεσης, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δεν υπάρχει κάποια μακροπρόθεσμη λύση εάν δεν δώσουμε οικονομικές ευκαιρίες και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης ε, στους νέους. Γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός παράγοντας στις χώρες της γειτονίας μας. Και ήθελα να τονίσω ότι όταν μιλάμε για την ασφάλεια εντός της Ευρώπης δεν υπάρχει πιθανότητα να εξετάσουμε την ασφάλεια μας χωρίς να εξετάσουμε και τις χώρες της γειτονίας μας. Ακριβώς γι' αυτό τονίζουμε τις εταιρικέ σχέσεις μας με τις χώρες της περιοχής και εξετάζουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας στην πολιτική συνεργασία μας με τις χώρες ε, της Μέσης Ανατολής. Ε, μόλις κατέβηκα από το αεροπλάνο επέστρεψα από τη Ιορδανία. Πραγματοποιούμε διάλογο και είναι ένα από τα παραδείγματα των περιπτώσεων όπου προσπαθούμε να έχουμε εταιρική σχέση με χώρες της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την εταιρική αυτή σχέση για ενίσχυση ε, της ανταπόκρισης ε, των, ε, απέναντι στις απειλές, Έχουμε εμπειρογνώμονες σε 9 από τις 10 αποστολές μας ε, στην περιοχή αυτή Έχουμε εκτεταμένους ε, διαλόγους ασφαλείας, ε, προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα τις χώρες της περιοχής και πώς μπορούμε να μάθουμε από αυτές. Μερικά από τα κρίσιμα ζητήματα έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού και την αντιμετώπιση των ιδεολογιών που οδηγούν στην ριζοσπαστικοποίηση. Επίσης συνεργαζόμαστε με ε, τις κοινότητες των ανθρώπων για να δούμε τι οδηγεί τον κόσμο στην ε, ριζοσπαστικοποίηση. Επίσης ε, προσπαθούμε να ανακόψουμε το ρεύμα των αλλοταπών πολεμιστών. 5.000 Ευρωπαίοι συμμετέχουν στις συγκρούσεις. Ε, δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε τα μέσα μας ε, με μια συνολική οπτική. Σημαντικό θέμα είναι επίσης η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Όπως σας είπα, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε τις ε, σχέσεις μας με τις χώρες της περιοχής. Όπως είπα στην αρχή της ε, παρέμβασής μου, υπάρχουν ε, πολλοί τρόποι να εξετάσουμε το θέμα της ασφάλειας. Ε, επικεντρώθηκα στο θέμα της τρομοκρατίας και της αιτίες της. Επίσης ανέφερα την οικονομική και κοινωνική διάσταση, ανέφερα και την πολιτική δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πολλά όσον αφορά την ε, ενίσχυση της ασφάλειας εντός της Ευρώπης. Για παράδειγμα, έχουμε την οδηγία για τα πυροβόλα όπλα για να αποφύγουμε τα πυροβόλα όπλα να πέφτουν σε λάθος χέρια. Επίσης, γίνονται προσπάθειες για την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και την αύξηση της διαλειτουργικότητας ανάμεσα στις διάφορες βάσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, αναγνωρίζουμε τα πλαστά διαβατήρια που χρησιμοποιούνται από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τρομοκρατικές ανέργειες. Αυτές λοιπόν είναι πτυχές που πολύ ευχαρίστω θα συζητήσω περαιτέρω μαζί σας. thank you very Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Κύριε Μπεναμούρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. έχω φέρει κάποιες διαφάνειες και σα ευχαριστώ που με προσκαλέσατε για να μιλήσω για τη Συρία. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν και να δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Συρία. Η πρώτη διαφάνεια. Βλέπετε την ιστορία των ΕΕ Συρίας, τι γίνεται με τη χρηματοδότηση 95.003 βάσει των εγγράφων της Κομισιόν. Θα δείτε ότι κάθε φορά που υπήρχε ένταση μεταξύ Συρίας και Ένωσης λάμβανε περισσότερα κονδύλια το καθεστώς Ασάντ μετά την κρίση. Όταν πέθανε ο πατέρας, ο Χαφές Ασάντ το 2000 είχαμε πολλές ελπίδες στην αποθέσει τον Μπασάρ Λασάντ και υπήρχε αισιοδοξία και μας απογοήτευσε και το 2004 και 2005 που δεν εφάρμοσε τις μεταρρυθμίσεις που νομίζαμε θα εφάρμοζε. Είχαμε και, το, και την δολοφονία του Ραρίφ Καδί από τις συριακές μυστικές υπηρεσίες. Το 2005 λοιπόν είχαμε μια πτώση. Μετά το 8 είχαμε μια αύξηση και το 9 και μια πτώση πάλι σήμερα μετά από τις δολοφονίες που διέπραξε το καθεστώς Ασάντ. Βάσει αυτών λοιπόν των στοιχείων να αναφέρω το γεγονό ότι βρήκα μια έκθεση Γενάρη 10 του Κοινοβουλίου, ίσως να ήσασταν τότε κάποιοι από εσά μέλη που ανέφερε αυτή την ε, έλλειψη συνέπειας μετά από επίσκεψη στην περιοχή και λέει η έκθεση που έχω εδώ μπροστά μου ότι τα κονδύλια για πολιτικές μεταρρυθμίσεις ε, υποχωρούν ενώ αυξάνονται αυτά για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Το λέγεται κοινοβούλιο. Δεν μπορούσε λοιπόν να έχει την κατάλληλη στάση ή παρά την αλλαγή των μεθόδων και της τάσης του Ασάντ. Επόμενη διαφάνεια. Διαφάνεια που έφτιαξα μαζί με τους αδέλφους από το Βεφημάτε στο κέντρο και εδώ βλέπουμε ακριβώς το πώς διοργάνεται η παρουσία της Ένωσης στη Συρία. Ίσως θα παρατηρήσετε κάτι βλέποντας αυτό το γράφημα, κάτι το οποίο εντυπωσιάζει. Λείπει εδώ παίκτη, το CSDP. Το CSDP δηλαδή η ασφάλεια και η άμυνα απουσιάζει από εδώ. Ντεύκο, η ΕΚΟ και άλλη μία για γενική της εδώ πρωτοστατούν με το συνδεσμό της υπηρεσία εξωτερική δράση. Αλλά ο στόχο εδώ είναι κυρίω βοήθεια για την ανάπτυξη. Νομίζω ότι αυτό αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο έχει δομηθεί ο προπολογισμό τη Ένωση. Μόνο 4% δηλαδή αφορά τα δικά θέματα, ασφάλεια κλπ. Και 30-35% αφορούν άλλε δράσει τη ΕΚΟ και τη ΤΕΦΚΟ. Αυτό που ονομάσαμε ως δευτερεύουσα τόσο παρέμβαση που έχει επιπτώσεις αλλά επιπτώσει που θα θέλαμε μια, πολιτική, μια πραγματική πολιτική παράδοση να έχει. Επόμενη διαφάνεια, τι κάνουμε εδώ. Όπω λέγαμε, μετά από πέντε χρόνια βοηθείς για την ανάπτυξη για τη Συρία. Μιλάμε για 5 έξι νομίζω τώρα, 6 δις ευρώ για τη Συρία και τις γειτονικές χώρες, δηλαδή Λίβανο, Ιορδανία, και η Τουρκία. Δεν περιλαμβάνει αυτό τη συμφωνία που είχαμε πρόσφατα με την Τουρκία. Και βλέπουμε στη διαφάνεια ότι τα περισσότερα χρήματα προέρχονται από τους Ευρωπαίους φορολογωμένους, κυρίως Γερμανία. Μετά τις, τη διάσκεψη του Λονδίνου, αλλά και εργαλεία της Κομισιόν και ΕΙΠΑ, έχουν σοβαρή παρουσία. Και παρατηρούμε επίσης ότι οι χώρες της μέση Ανατολή είναι αρκετά χαμηλά. Έχουν χαμηλή δηλαδή παρουσία σε αυτό το γράφημα. τα πράγματα από αυτή τη σκοπιακή και πέρσι και συνεχίζουν να είναι και σήμερα. Επόμενη διαφάνεια. Το 2013 απάντηση σε αυτά που συνέβαιναν στη Μέση Ανατολή έχουν σημειωθεί, μάλλον επιτευχθεί διάφορα μέχρι τώρα από τότε γιατί είχαμε την υποχώρηση ας πούμε του Ισλαμικού κράτους σε πιο ε, εσωτερικέ περιοχές έχουμε την κατάσταση στην Τουρκία έχουμε τις εξελίξεις που αφορούν ε, Ιορδανία και Λίβανο και έχουμε και την ΕΚΟ που είχε αναλάβει για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη Συρία. Έχουμε λοιπόν μια οργάνωση επίπεδο ενωση. που διοργάνωνε την, το συντονισμό όλης της παρουσίας και της συμβολής της Ένωσης. Πώς δεν ξέρω αν θέλετε να τον βαθύνω αυτό στις επόμενες διαφάνειες. Πάντως, όπως λέγαμε, αυτή η βοήθεια, η παροχή της δεν είναι και τόσο ορατή, γιατί αυτά τα κονδύλια δαπανώνται μέσω κυρίως του ΟΗΕ. Επόμενη διαφάνεια. Τελευταία διαφάνεια που σας δείχνει την κατάσταση στο Χαλέπι. Εδώ βλέπουμε την πρόοδο των στρατιωτικών δυνάμεων του Βασάρα Λασάντ δεν θα μιλήσω βέβαια για τη θεωρική κατάσταση, θα διαβάσετε στον τύπο, αλλά να σας πω εδώ τι σημαίνει αυτό για μας, για τους Ευρωπαίους. Αυτό σημαίνει ότι πριν είχαμε μια προσέγγιση 50-50 στη Συρία, δηλαδή 50% τη βοήθεια πήγαινε στη Δαμασκό και 50% στο Βορρά. Είχαμε όμως, έχουμε όμω σταματήσει αυτή την προσέγγιση και θα πρέπει να συζητήσουμε και συζητήσαμε τον με το του Δαμασκού πώς θα διοχετεύεται στη Συρία αυτή η βοήθεια, αλλιώ δεν θα δοθεί. Και αυτό το κύριο το θέμα θα πρέπει να συζητήσουμε εδώ. Δηλαδή τις αρνητικές επιπτώσεις και τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής βοήθειας γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ή κάποιοι από τους συζητητές που ήρθαν σα πούν ότι κάποια από αυτή τη βοήθεια πήγε στο Ισλαμικό κράτος ότι κάποια από αυτή τη βοήθεια πήγε στον και στα περιοχές που, όπου έχει κυριαρχήσει. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις περιοχές που έχει κτίσει το καθεστώς του Πασαρασάρ. Παρέχει κονδύλια βέβαια ο ΙΕ για αυτούς που χρειάζονται βοήθεια. Υπάρχουν όμως και κονδύλια τα οποία χρησιμοποιούνται για να σταθεροποιηθούν τα κεκτημένα του καθεστώτος του ασάδ ή του Ισλαμικού κράτους. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να δούμε εδώ σε επίπεδο λεπτομέρειες τι συμβαίνει. Εγώ δεν είδα κάτι παρόλο που το έψαξα. Και ξέρω ότι υπάρχουν ευαισθησίε, και ότι θα πρέπει να πάρουμε σκληρέ αποφάσεις, αλλά εδώ ακριβώς η Ευρώπη πρέπει να ηγείται. Αυτό το οφείλουμε στους φορολογούμενου και στους εαυτούς μας. Δηλαδή να έχουμε ένα σαφή ορισμό που πηγαίνει ακριβώ η βοήθειά μας. Αυτά από μένα και σα ευχαριστώ που με ακούσατε. Είμαι εδώ και για ερωτήσει που θα είχατε όσον αφορά αυτή την βοήθεια για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ και πάλι. Okay. Ωραία. Παρακαλώ τα μέλη που επιθυμούν το λόγο να σηκώσουν το χέρι για να καταγραφούν στο κατάλογο των ομιλητών. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που λέτε για το ποια είναι η πραγματική αιτία της σύγκρουσης. Και πρέπει να πάμε πίσω στις ρίζες αυτή της Συριακή σύγκρουσης. Και αυτό είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έχει αγνοήσει, δεν έχει κάνει, γιατί βέβαια υπήρξαν διαμαρτυρίες. Αν είχε πιο ενεργό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από πέντε χρόνια στην αρχή της κρίσης αυτής, τότε ίσω η κατάσταση να μην είχε φτάσει στα άκρα όπως έχει φτάσει τώρα. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αλλαγή της κατάστασης ήταν δευτερεύον. Ο ρόλος μας ήταν να είμαστε ο καλός Σαμαρίτης, χωρίς να προλαμβάνουμε τίποτα, χωρίς να λύνουμε τίποτα, να εφιστάμεθα τις συνέπειες και να αναλαμβάνουμε τις συνέπειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έμεινε στην πάντα, ως παρατηρητής πάντα. Έπειτα, το θέμα αυτό του πληθυσμού που φεύγει και που τον σπρώχνει έξω από τη χώρα ο ίδιος ο Ασάντ. Υπάρχει συνύπαρξη ανάμεσα στον Ασάντ, τη δικτατορία του Ασάντ και το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Γιατί κάποιος από τους εμπειρογνώμονες μας είπε πριν από μερικές εβδομάδες ότι το πετρέλαιο από τα κατεχόμενα από το Ισλαμικό κράτος εδάφη στέλνεται με αγωγούς στα κομμάτια της Συρίας που ελέγχει ο Ασάντ και και οι δύο πλευρές και το Ισλαμικό κράτος δηλαδή και ο Ασάντ αποφελούνται. Πώς εκτιμάτε την αλυσίδα των ε, συμμάχων Ρωσία, Ασάντ, Ιράν, που το Ιράν ενισχύθηκε μετά από την πρόσφατη πυρηνική συμφωνία. Και ο κουρδικός παράγοντας τι ρόλο παίζει σε αυτή την κατάσταση. Οι Κούρδοι έχουν κατακαιρματιστεί, αλλά έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Παρακαλώ. Η Ευρώπη εξαφανίστηκε από τη Μέση Ανατολή. Τώρα απλώς είμαστε πάροχοι ανθρωπιστικής βοήθειας. Άμυνα εξωτερική πολιτική ανύπαρκτη. Από την αρχή ανύπαρκτη. Όταν οι αντιστασιακοί επαναστάτες, όπως θέλετε τους λέτε, άρχισαν, είπαμε τις ίδιες ανοησίες που είπαμε και την εποχή της Βοσνίας και Ερσεγοβίνης, ότι δεν θέλουμε να εθαρρύνουμε τη βία. Οπότε κάθε είδους καταστροφή, ε, βιασμοί, δολοφονίες, ε, μαζικές ε, απαγωγές, όλα έγιναν. Γιατί δεν στηρίξαμε αρκετά τα πράγματα ώστε να ρίξουμε τον Ασάντα. Δεν στηρίξαμε τον Ασάντ βέβαια, δεν στηρίξαμε όμως και την ανταπολίτευση για να γίνει αρκετά ισχυρή ώστε να φύγει ο Ασάντ όταν άρχισε ο στρατός του να διαλύεται. Και εδώ φτάσαμε σήμερα και διάβασα στον Ισπανικό τύπο μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Επισκόπου του Αλέπου. Λέει ότι ο μισός ε, πληθυσμός της Συρίας θα στηρίξει τον Ασάντ ακόμα και αν τον μισεί γιατί βρίσκεται μεταξύ διπλών ε, πυρών σε μια κατάσταση γενοκτονίας. Έχουμε λοιπόν τον Ασάντα από τη μία μεριά, αλλά είναι η μόνη δυνατή απάντηση απέναντι στο φανταματαλισμό μεταξύ άλλων και της Αλκαΐντα και του Ντάς που έτσι καλλιώς είναι διακλαδώσεις του ίδιου βασικού κορμού. Τι πετύχαμε? Να βάλουμε τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή, νομίζοντας ότι δεν υπήρχε η Ρωσία. Και σήμερα διαπιστώνουμε ότι πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία, που είναι γειτονική χώρα, και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί η Ευρώπη δεν κατάφερε να προφέρει ούτε μία λέξη σε ένα πόλεμο, ο οποίος συνεχίζεται πέντε χρόνια τώρα. Και ανησυχούμε για τους πρόσφυγες, γιατί δημιουργούν προβλήματα στην Νότια Ευρώπη όχι γιατί έχουμε τρυφερή καρδιά. Είναι αξιοθρύνητη η κατάσταση των ε, προσφύγων για χρόνια. Φωτογραφίες μόνο όπως το Αιλάν που βρέθηκε νεκρός στις ακτές της Τουρκίας. Αν κάτι ενοχλεί το γεύμα μας, την ώρα που τρώμε και βλέπουμε τις ειδήσει ε, στην τηλεόραση, ε, αυτό μόνο μας παρακουνάει κάπως. Τίποτα άλλο. Και βάζουμε και το Ιράν ε, με δύναμη στην περιοχή όπως δεν ήταν ποτέ. Το Ιράν και η Ρωσία θα αποτελέσουν τους σταθεροποιητικούς παράγοντες στη Συρία και το Ιράκ. Χωρίς το Ιράν σήμερα η Ντάς θα στη Βαγδάτη, το Ισλαμικό κράτος. Οπότε τι λέμε τώρα. Πού είναι η Ευρώπη. Εγώ δεν τη βλέπω. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Κούσο έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα εγώ από την πλευρά μου να επικεντρωθούμε κάπως περισσότερο μια στιγμή. Μια στιγμή να βάλει ο κόσμος τα ακουστικά του. Περιμένετε, λέει ο Πρόεδρος. Ωραία, έλεγα λοιπόν ότι θα ήθελα να επικεντρωθούμε κάπως περισσότερο στο θέμα της ασφάλειας. Όταν αναφερθήκατε στη χρηματοδότηση για παράδειγμα, γιατί ακριβώς με αυτό πρέπει να τα βάλουμε. Η εσωτερική ασφάλεια είναι όπως και η εξωτερική ασφάλεια. Αυτό που ονομάζεται Ισλαμικό κράτος, Καλυφάτο, είναι εκεί όπου έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι τζιχαντιστές και τώρα μας έρχεται σαν μπούμεραγκ σε εμά σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους λέμε βαρβάρους. Ωραία, πώς όμως θα καταφέρουμε να πνίξουμε αυτό το φαινόμενο αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Τώρα άκουσα, αν είχε και λόγια εδώ πέρα από τους ομιλητές, αναφερθήκατε στην προπαγάνδα, μετά μιλήσατε για το Hollywood και ότι τα αναλάβαμε όλα αυτά και ο Ασάντ είπατε ότι είναι ο μόνος υπεύθυνο για τους χιλιάδες νεκρούς. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό. Όταν λέτε ότι την κατάπαυση πυρός την πέτυχε το Μετροπαθές Κέντρο, εγώ δεν ξέρω που βρίσκεται αυτό το Μετροπαθές Κέντρο, εγώ ξέρω ότι μια συμμαχία κατά του Ισλαμικού κράτους εδώ και ένα χρόνο βομβαρδίζει και δεν προχωράει τίποτα. Τίποτα. Επιτόπου τίποτα δεν αλλάζει, τίποτα δεν γίνεται. Και γιατί, γιατί το ξέρουν όλοι. Γιατί όταν συνδυάζεται οι αεροπορικές δυνάμεις χωρίς ε, στο έδαφος ε, δυνάμεις δεν γίνεται τίποτα. Ενώ η Ρωσία είχε και την αεροπορική κάλυψη αλλά είχε στρατεύματα και ε, κάτω. Οπότε το να μιλάμε για αυτό το μετροπεθέ κέντρο, εγώ δεν ξέρω που το βλέπετε εσείς αυτό. Τώρα η, Ρωσία δεν τα έβαλε με το Ισλαμικό κράτος και δεν τέλειωσε με τη σύγκρουση αυτή. Πάλι μακιανιστικό μου φαίνεται αυτό που λέτε, ότι η Ρωσία είναι όλα τα κακά. Εντάξει, φυσικά και έχει τα δικά της τα συμφέροντα, πολύ θα ήθελε να έχει ταρτούς, να έχει διέξοδο στη θάλασσα, αλλά δεν θα πρέπει να λέμε ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα και στη Ρωσία το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Είναι δίπλα στα σύνορά της. Ανεξάρτητα τώρα από το τι νομίζει ο καθένας, για να υπάρξει μια λύση, φυσικά και πρέπει να είναι παρούσα και η Συριακή κυβέρνηση. Πάντα στηρίζαμε τον Ταμιστούρο των ειδικό απεσταλμένο και η Ισπανία δυστυχώς και αυτή θα συμμετάσχει θα στηρίξει τις συνομιλίες για την ειρήνευση στη Συρία, ελπίζοντας ότι δεν θα έχουμε τέτοια αποτελέσματα όπως είχαμε και στο Ιράκ ή όπως έχουμε στη Λιβύη. Δεν θέλουμε να γίνει το ίδιο και στη Συρία, ένα αποτυχημένο κράτος. Θα ήθελα επίσης να αναφερθείτε λίγο και για το ρόλο των χωρών του κόλπου. Η Τουρκία τι ρόλο παίζει στη χρηματοδότηση του Ισλαμικού κράτους. Ή από την άλλη μεριά. Είχαμε εδώ τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Ιράκ που μίλησε για το πετρέλαιο και για την ε, μεταφορά του από το Ισλαμικό κράτος αλλού προς αλλού. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Κύριε Βαλέρο, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιος από εσά μίλησε για μία λύση με επικεφαλή στη Συρία. Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις αυτές και πολλοί από αυτούς καθορίζουν ποιοι θα συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και ποιοι όχι. Αναρωτιέμαι λοιπόν είναι βιώσιμη μία λύση με επικεφαλή στη Συρία ή θα καθοδηγηθεί από αλλού. και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορούμε να κάνουμε. Η ε, κυρία Ζενή μίλησε για τους 5.000 αλλοδαπούς πολεμιστές. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει όμως να κάνουμε και περισσότερα όσον αφορά την διπλωματία, την αναπτυξιακή βοήθεια κλπ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο μεγαλύτερος χορηγός σε όλον τον κόσμο να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας για να βοηθήσει τους ανθρώπους της περιοχής αυτής που υποφέρουν. Δεν ξέρω αν κατάλαβα σωστά. Νομίζω, κύριε Βενχαμού, ότι αναφερθήκατε και στην ε, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και τις προσπάθειες που κάνουμε. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει στρατιωτική επέμβαση, διότι γνωρίζετε ότι οι ε, Ηνωμένε Πολιτείε και οι Κούρδοι καταπολεμούν ε, το ISIS, οι Τούρκοι καταπολεμούν τους Κούρδους, ε, ο Ασάντ πολεμάει ενάντια στην αντιπολίτευση. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε στρατιωτική επέμβαση και αν είναι πού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Actually, I would follow Ο επόμενος ομιλητής θα συμφωνήσω με τις ερωτήσεις σας, ε, ιδιαίτερα προς ε, τον πρώτο ομιλητή, διότι είπατε όχι μόνο ότι είναι προβλέψιμο, αλλά ότι είχε προβλεφθεί κιόλα. Πιστεύετε ότι πρέπει να μάθουμε από αυτά που έκανε η Ρωσία. Η Ρωσία έκανε σταθερική παρέμβαση και επέμβαση και άλλαξε το παιχνίδι. Όλα ξεκίνησαν βέβαια με τον Ομπάμα και τις κόκκινες γραμμές του. Τι συζητάμε εδώ. Να παρέχουμε απλά ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς πολιτική βούληση και χωρίς στρατιωτική δύναμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαφοζέρ. ήταν ευγενικοί οι συνάδελφοι στι κριτικέ του. Όπω ο φίλος Τανζόν, θα μπορούσα να φύγει κι εγώ. Κάνοντα έτσι μια χειρονομία. Ο γνώστη, όπω ο συνάδελφος Τανζόν. Εγώ δεν ήμουν ε, διευθυντή γραφείου του υπευθύνου πληροφοριών, αλλά για χρόνια ήμουν στον ΩΣΑ, ήμουν και αντιπρόεδρος η πρώτη δηλαδή η Ευρωπαϊκή ΜΚΟ που παρανέβει στη Συρία. Έχω λοιπόν κάποια σχέση με αυτό το μέρος και ξέρω δύο πράγματα για την νομιμότητα ή όχι του Ασάντ, τουλάχιστον όσον αφορά τι χριστιανικέ μειονότητε, για τι οποίε όμω εμεί δεν παρεμβαίνουμε. Εμεί ξέρετε ότι παρεμβαίνουμε για όλου. Και είμαστε ανοιχτοί προ όλου. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια φάση αποσταθεροποίηση ενό συστήματο. Το όταν και στο Ιράκ. Υπάρχουν βεβαίω ευθύνε του Σαντάμ ή στην Λιβύη του Καντάφη, όπως και στη Συρία. Όταν όμως μια εξωτερική δύναμη κρίνει ότι η τάδε η δυνα κυβέρνηση δεν είναι βιώσιμη και προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει μέσω πολέμου μόλις τις συνέπειες που έχει γεωπολιτικά αυτό, τότε είμαστε εκτός διεθνούς δικαίου, είμαστε εκτός κανόνων πάνω στους οποίους πράγματι βασίζεται και στηρίζεται η ειρήνη. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε μόνο με τα Ηνωμένα Έθνη. Πραγματικά είμαι αγανακτισμένος με αυτά που ακούω από εσά. Όταν βάζετε στο ίδιο επίπεδο μια κυβέρνηση, παρόλα αυτά που είναι νόμιμη και που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ και τη βάζετε στο ίδιο επίπεδο με το Ισλαμικό κράτος. Είναι απαράδεκτο αυτό που λέτε. Δεν θα μπορούσατε, θα έπρεπε να έχετε πρόσβαση εδώ στο Κοινοβούλιο να λέτε τέτοια πράγματα. Είμαι αγανακτισμένο. είμαι αγανακτισμένο. Κυρία Πρόεδρε, σα παρακαλώ πολύ μη φωνάζετε λέει η Πρόεδρε, σας παρακαλώ, σα ακούμε. Είμαι αγανακτυπισμένος λοιπόν, σκανδαλώδια αυτά που λέτε. Όταν λέτε ότι η Ρωσία παρενέβη υπέρ του Ασάτ να δεχτείτε τουλάχιστον ε, το εξή, επειδή έχω επαφές και με τη Ρωσία. Η Ρωσία ανησυχεί για την διεθνή τρομοκρατία από την οποία έχει υποφέρει. Ανησυχεί λοιπόν για αυτό το φαινόμενο και με το Ισλαμικό κράτος και τη διεθνή τρομοκρατία, ε, ε, τρομοκρατία που είχε χειραγωγηθεί. Και συμφωνώ εδώ και από ό,τι είπα Υπάρχει εδώ, εδώ, λοιπόν εδώ ένας πραγματικός κίνδυνος. Έπρεπε να σταματήσει η επέκταση του Ισλαμικού κράτους. Να σας πω λοιπόν για αυτά που λέτε ότι ο φίλος μου εδώ που ξέρει πολύ καλά την κατάσταση επειδή ήταν υπεύθυνο ε, των πληροφοριών και όλοι αυτοί που έχουν σήμερα ευθύνε, τι ιστορίε και αυτά που λέτε δεν τα πιστεύουμε. Ήταν καθαρά ιδεολογικά, ιδεολειπτικά. Δεν σα πιστεύουμε ούτε καν στη Γαλλία, ούτε καν στο Παρίσι, ούτε καν οι μετριοπαθεί. Και με του αφού μουσουλμάνου που χειραγούν την ε, αντιπολίτευση, με την Τουρκία, με το Κατάρ από πίσω. Πώς τολμάτε, πώς τολμάτε σήμερα να, να έρχεστε εδώ να μας λέτε τέτοια πράγματα. Δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε να καθόλου από αξιοπρέπεια. Τροπή σας. Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας δώσω το λόγο στους υπόλοιπους σε λίγο. Θα ήθελα μόνο να απαντήσω στον κ. Σαχάουζερ. Δεν χρειάζεται να φωνάζετε. Και βεβαίω δεν χρειάζεται να μας κατηγορείτε. Με αυτά που είπατε. Για την επιλογή των ε, υπερογνωμών Αυτοί επιλέχθηκαν από τους συντονιστές. Συμφώνησαν οι συντονιστές γι' αυτό. Και για διάφορους λόγους η πρόταση μου δεν ληφθεί υπόψη. Πρέπει όμως να παραδεχτώ ότι αυτή η επιλογή προκεκλημένων και εισηγητών από τους ε, συντονιστές ε, με βρίσκει σύμφωνη και νομίζω ότι είναι σωστή. Παρόλο που πράγματι δεν αποτέλεσε δική μου απόφαση, γιατί έχουμε εδώ μια ακρόαση. Και υπάρχει το έθιμο εδώ στο σώμα μας, οι συντονιστές, να λαμβάνουν τι αποφάσεις για αυτά τα θέματα. Τρίσκο. Ε, Pani e, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να αναφερθώ σε αυτά που ακούσαμε ακριβώς πριν, γιατί έχω διάφορα σχόλια. Κανείς δεν πιστεύει, κανείς δεν είναι πεπισμένος για το ποια είναι η αλήθεια. Εγώ πιστεύω αυτά που είπατε, αυτά που λέτε. Εγώ πιστεύω ότι η περιγραφή που κάνατε της κατάστασης είναι ορθή. Οπότε διαμαρτύρομαι για αυτά που είπε ο κ. πριν από λίγο. Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι η κατάσταση όντως είναι περίπλοκη. Και κανείς δεν μπορεί να πει ότι μπορεί να βρεθεί υπάρχει μια απλή λύση. Δεν υπάρχει. οποιαδήποτε πλευρά που έχει εμπλακεί η σύγκρουση έχει κάνει λάθη. Καμία δεν είναι εντελώς αθώα. Σήμερα όμως πρέπει να δράσουμε για να ελαχιστοποιήσουμε τα σφάλματα αυτά και να διασφαλίσουμε ότι τα θύματα είναι όσο γίνεται λιγότερα εξαιτίας των σφαλμάτων αυτών. Αλλά διαφωνώ πλήρως με αυτά που είπε ο συνάδελφος πριν. Εμένα με ικανοποιεί η παρουσίασή σας και ο τρόπος που παρουσιάζετε εσείς την κατάσταση. Και έτσι είμαστε πιο κοντά προς την λύση, πιστεύω, με αυτόν τον τρόπο. Ναι, εγώ τώρα. Πριν σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε, είναι η δικιά μου σειρά. Λέει πρόεδρος. Ναι, λοιπόν πιστεύω και εγώ ότι ήταν πολύ καλή η παρουσίασή σας και όντως μας φέρνει πιο κοντά σε μια πραγματική εκτίμηση της κατάστασης που σίγουρα είναι πολύ δύσκολη και πολύ θλιβερή. Αλλά γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και πρέπει να επιτρέπουμε πραγματική ανταλλαγή απόψεων. Ακόμα και τις απόψεις του κύριου Σαφχάουζε με τις οποίες εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα και σε τέτοιες φωνές να ακούγονται. Γιατί στο κάτω-κάτω αν οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται εδώ είναι γιατί κάποιοι τους ψήφισαν. Λοιπόν, τώρα, ε, με ενδιαφέρει πολύ η εκτίμηση που κάνετε όσον αφορά τη στατική αυτή του Ασάτ να κάνει τον κόσμο να φύγει από τη χώρα. Ο κύριος Χόικεν ήταν αυτός που μας παρουσίασε αυτή την άποψη. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Και ίσως έτσι μπορούμε να προβλέψουμε και τη συνέχεια. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να αναπτύξετε περισσότερο αυτή την ε, τοποθέτησή σας. Εγώ θυμάμαι πριν από τέσσερα χρόνια περίπου, νομίζω. Όταν μπορούσαμε να συζητήσουμε για το Νόμπελ προκειμένου να λυθεί η κατάσταση αυτή στη Συρία. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα ήταν τότε το θέμα των εξοπλισμών, των χημικών όπλων, αν υπήρχαν εκεί και πώς θα μπορούσαμε πολιτικά να λύσουμε την κατάσταση. Είπατε επίσης ότι αν αποσυρθεί ο Ασάντ θα καταλήξουμε σε μια παγωμένη σύγκρουση. Πιστεύετε ότι αυτός ήταν ο στόχος ε, του ενός παίκτη ή περισσότερων και τι θα γίνει στη συνέχεια. Και προς την κυρία Ζωέλ θέλω να ρωτήσω το Υπήρξαν κάποιες ενδείξεις για κατάχρηση ανθρωπιστικής βοήθειας ή ότι η ανθρωπιστική βοήθεια τέλο πάντων πήγαινε σε περιοχές που ελέγχονται από τον Ασάντ. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ώστε η ανθρωπιστική αυτή βοήθεια να φτάνει πιο ισορροπημένα γεωγραφικά τουλάχιστον στη χώρα ώστε να φτάνει σε περισσότερους ανθρώπους σε μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας των πολιτών στη Συρία. Τι προβλέπετε εσείς για την κατάσταση. Εκεί όπου υπάρχουν πάρα πολλοί Σύριοι πρόσφυγες στην Τουρκία, το Λίβανο, η Ορδανία. Ξέρω ότι η κατάσταση την Ιορδανία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πολύ δύσκολη ήδη όσον αφορά την ανθρωπιστική κρίση. Τι λέτε λοιπόν, τι θα έπρεπε να είναι το επόμενο βήμα μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Με την ίδια σειρά νομίζω. Ε? Τι λέτε. Ο κύριος Χόκα για μισός επειδή πρέπει να φύγει και νωρίτερα. Ε? Πρώτος εσείς λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπώ τη δημοκρατία. Μ' αρέσουν και οι διαφωνίες. Θα ευχόμουν να ήταν εδώ ο Ευρωβουλευτής ε, να το ακούσει αυτό. Είμαι εμπειρογνώμων, κάνω έρευνες, ε, δεν έχω πολιτικό θεματολόγιο. Εξετάζω πώς έχουν τα πράγματα και θα ήθελα να διαβεβαιώσω σε όλους εδώ ότι δεν ε, έχω άλλα κίνητρα. Η πραγματικότητα σήμερα στην Συρία είναι ότι οι περισσότεροι Ε, θάνατοι τυχαίνει να είναι φτωχοί ε, Σύριοι που είναι Άραβες Σουνίτες. Ε, θα πρέπει βέβαια να εξετάσουμε και την κατάσταση των μειονοτήτων συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών στη Συρία. Αλλά το να μεγεθύνουμε το θέμα τους σε σχέση με άλλους τους κάνει πιο ευάλωτους σε αντίπεινα. Υπάρχει κίνδυνος ε, το καθεστώς ε, Ασάντ να τους κρατήσει ομήρους, ακριβώς τους ανθρώπους ε, που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που αρνούνται την εξίσωση ανάμεσα σε αυτούς και το καθεστώς και δεν θα πρέπει να πέσουμε εδώ στη Δύση στην παγίδα αυτή. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε την ε, βιότητα του καθεστώτος ε, Ασάντ επειδή μας ενδιαφέρουν οι μειονότητες. Θα πρέπει να εξετάσουμε όλη την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ε, μαζικές δολοφονίες έχουν στόχο τους φτωχούς Σουνίτες στη Συρία. Να είμαι σαφής λοιπόν όσον αφορά το θέμα αυτό. Το θέμα των μειονοτήτων είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, επίμαχο είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πολλούς. Εμένα σίγουρα σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αλλά να προσέξουμε να αποφύγουμε την ε, εξίσωση αυτή διότι έτσι θέτουμε σε κίνδυνο πολλούς ανθρώπους. Θα ήθελα η Ρωσία να έχει στραφεί περισσότερο κατά ε, του ISIS, του Ισλαμικού κράτους εξετάζουμε τα στοιχεία αλλά ε, μας δείχνουν τα στοιχεία αυτά ότι το 15% των ρωσικών επιθέσεων είχαν στόχο το Ισλαμικό κράτος. Οι κυβερνήσει σας φαίνεται επίσης να συμφωνούν με, με αυτόν τον υπολογισμό. Δεν το αμφισβητούν πολύ αυτό λοιπόν, αλλά ένα άλλο θέμα που τέθηκε έχει να κάνει με την ε, πολυμορφία των επαναστατικών ομάδων εντός της Συρίας και καταλαβαίνω ε, γιατί όλο αυτό προκαλεί σύγχυση. Δεν είναι όλοι τσιχαντιστές. Άκουσα να αναφέρεται το Ζήσελ Ισλάμ, ε, είναι ριζοσπαστικές ομάδες Ισλαμιστών, δεν είναι όμως τσιχαντιστές. Είναι δεν είναι εξτρεμιστές, είναι ριζοσπαστικοί, θα πρέπει να τους περιορίσουμε πολιτικά δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υποστήριξη, αλλά αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του πληθυσμού. Χωρίς αυτούς ε, θα είναι αδύνατο να πετύχουμε τη σταθερότητα που θέλουμε. Ε, το Ζάμπατ Νούσρα, ε, η ISIS και άλλοι είναι καθαρά ομάδες τσιχαντιστών. Ποια ομάδα νομίζετε ότι έχει περισσότερο αίμα στον αγώνα κατά της ISIS, η Αχαρισάμ το 2014. Λόγω των όσων συνέβησαν, από το Σεπτέμβριο του 2014 και μετά. Θυμόμαστε τις τεράστιες θυσίες, τις ε, θυσίες των Κούρδων, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ε, το Ισλαμικό κράτος εκδιώχθηκε από την ε, Βόρεια Συρία μέσα σε λίγες εβδομάδες από 3,5 περιφέρειες εκδιώχθηκε χωρίς δυτική βοήθεια ή πληροφορίες από τη Δύση. Πού έχουν οι Κούρδοι σήμερα. Θα ήθελα να καταλάβετε τη δυναμική. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι η, ε, ο θρίαμβος ε, της μιας ομάδας ε, πάνω στους άλλους. Δεν υπάρχει στρατιωτική νίκη για κανέναν στη Συρία, ούτε για τους επαναστάτες στόχος δεν ήταν ποτέ οι επαναστάτες να ε, κατέχουν την Δαμασκό. Το Χαλέπι ήδη έχει καταστραφεί και οι επαναστάτες ε, ήδη έκαναν το λάθος να προσπαθήσουν να καταλάβουν αυτήν την μεγαλύτερη πόλη ε, και πληρώνουν το τίμημα όπως και οι απλοί πολίτες πληρώνουν το τίμημα. Το θέμα είναι λοιπόν τους επαναστάτες να τους περιορίσουμε, να ε, τους φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ο Ασάντ να καταλάβει ότι ε, ο χρόνος που θα παραμείνει στην εξουσία δεν είναι οριστός. Δεν, δεν θα παραμείνει για πάντα στην εξουσία. Δεν υπάρχει όμως μια εύκολη πολιτική λύση που κατάλαβε η Ρωσία. Η Ρωσία διαμόρφωσε το πεδίο μάχης, ε, την διπλωματία με χαμηλό κόστος. Πιστεύω λοιπόν ε, εγώ ότι οι χώρες της Δύσης και οι σύμμαχοί τους είχαν ε, την ευκαιρία να το κάνουν αυτό. Όχι. Πιο εύκολο είναι να υποστηρίξει κανείς ε, μια υπάρχουσα κυβέρνηση με πρωτεύουσα από την επανάσταση που θέλει να τα ανατρέψει. Η μόνη χρονική στιγμή που θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι τέτοιο ήταν τον Οκτώβριο-Σεπτέμβριο του 2013 όπου υπήρχε σαφής λογική, υπήρχε κόκκινη γραμμή. Ε, δεν δόθηκε συνέχεια όμως ε, ο Ασάντ. Εποφελήθηκε από το ψήφισμα για τα χημικά όπλα. Και τέλος, ε, όσον αφορά το θέμα που θίξατε, δύο παρατηρήσεις ακόμα. Η στρατηγική Ε, για τον ε, πληθυσμό. Δεν είναι πολύ επίμαχο το θέμα αυτό μεταξύ των εμπειρογνωμών. Υπάρχουν ε, πληθυσμοί που ο Ασάντ θεωρεί κατανοητό αυτό ότι είναι άπιστη απέναντί του. και με πολιτικούς και οικονομικούς τρόπους προσπαθεί να τους καταπολεμήσει. Οι περισσότεροι από αυτοί είναι πρόσφυγες σήμερα στην Τουρκία, στο Λίβανο, στη Ιορδανία δεν απασχολεί... Δεν απασχολούν όμως αυτοί τον Ασάντ, αλλά η Δυτική Συρία, όπου βρίσκονται τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, οι υποδομές, ε, τα τρόφιμα κλπ. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να οδηγήσουν στο απόλυτο χάος. Εμείς μιλάμε για τον αγώνα κατά του Ισλαμικού κράτους, αλλά το πρόβλημα είναι ποιο θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Εάν δεν λάβουμε υπόψη μα την πολιτική της Ρωσίας, οι Κούρδοι μπορεί να καταλάβουν τη ράκα, αλλά θέλουν να καταλάβουν τη ράκα, όχι. Θέλουν να δημιουργήσουν μια βιώσιμη οντότητα, κάτι που έχει νόημα από τη δική τους πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν έχουμε τοπικούς αραβικούς παράγοντες ε, που να είναι κατά του Ισλαμικού κράτους, μπορεί η Ιράκα να ερημώσει τελείως. Και η τελευταία μου παρατήρηση είναι... Θα πρέπει να ξεφύγουμε από την ιδέα ότι έχουμε την επιλογή ανάμεσα στον Ασάντ και το Ισλαμικό κράτος ή ότι ο διαχωρισμός είναι ανάμεσα στον Ασάντ και ένας γενικός εξτρεμισμός. Δεν είναι αυτή η επιλογή. Ε, υπάρχουν πολλοί διαχωρισμό ε, ικανοί ε, Σύριοι. Μερικοί από αυτούς βρίσκονται στην Γενέβη και ένα γενικος εξτρεμισμο δεν ειναι αυτη η επιλογη υπαρχουν πολλοι αξιοπρεπεις πολύ ικανοι συριοι μερικοι απο αυτού βρισκονται στην γενεβη και, συζητουν με ευρωπαιους υπουργού και αλλους για να βρουν εφαρμόσιμες λύσεις. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι εξίσου αφοσιωμένοι στον αγώνα κατά του Ισλαμικού κράτους όσο είναι και κατά του Ασάντ. Υπάρχουν μέρη του καθεστώτος ε, Ασάντ που θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος σε μιας ενδεχόμενης λύσης. Και αυτό το αναγνωρίζουν άνθρωποι της αντιπολίτευσης, αλλά πρόκειται για αναθεωρητισμό του χειροτέρου είδους να ε, υποτιμούμε τη σημασία των Ασάντ και ιδιαίτερα του Μπασάρα Ασάντ ε, στην σύγκρουση αυτή. Αυτό γίνεται στο όνομα της προστασίας ε, μειονοτήτων, ε, ε, διότι υποτίθεται ότι ο Ασάντ είναι κοσμικός. Δεν μπορώ ακριβώς να καταλάβω πώς ορίζεται αυτή η λέξη του κοσμικού κράτους ή του κοσμικού ατόμου στην Μέση Ανατολή, αλλά η Συρία δεν πρόκειται να σταθεροποιηθεί εάν επιτρέψουμε να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η εξίσωση στο μυαλό μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία τώρα. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Χοκέλια που συνέβαλε με τρόπο που συχνά λείπει από τις συζητήσεις μας για τη Συρία. Νομίζω ότι αυτά που είπατε είναι πάρα πολύ σωστά και πολύ σημαντικά επειδή η χάραξη πολιτικής από απόσταση χωρί κατανόηση τη περιπλοκότητα και των επιχειρημάτων των εμπλεκομένων και τη δυναμική και το γεγονό ότι δεν υπάρχουν άσπρες μαύρε λύσεις είναι βασική σημασία. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε περισσότερο και σε βάθος στη Συρία ποιοι είναι οι παίκτες, τι επιπτώσεις υπάρχουν, σε συνεργασία με διάφορους συνεργάτες που είχαμε παντού στη Συρία και τους προστηρίξαμε και από την υπηρεσία, από το γραφείο που δημιουργήσαμε στο Καζεντέ που ήταν πολύ ενεργό στην παροχή βοήθειας και στήριξης. Προσπαθήσαμε λοιπόν να καταλάβουμε και να αναλύσουμε την περιπλοκότητα της κατάστασης για να στηρίξουμε την διπλωματική μας προσπάθεια. Τώρα η Ένωση έκανε μια σαφή επιλογή για την υποστήριξη της διπλωματικής οδού με τον κύριο Μιστούρα τον ειδικό Εγώ είμαι υπεύθυνη και της μονάδας μεσολάβησης και ξέρουμε ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις το χειρότερο, η χειρότερη εξέλιξη είναι το να υπάρξει διάσπαση. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε στην ε, συνάντηση Γενέβης και στην υποστήριξη του κ. Δεμιστούρα. Αυτό είναι κεφαλαίο του σημασίας. Και θα έπρεπε η Ένωση να μην ακολουθήσει διαφορετική διαπραγματική οδό. Υπάρχουν τα σημεία Γενέβη που έχουν συμφωνηθεί, υπάρχει μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται και όλοι πρέπει να εμπλακούν μέσω διπλωματικών οδών στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας μεσολάβησης. Το ανθρωπιστικό ζήτημα είναι τεράστια δυσκολίας και έχει τεράστιες ανθρώπινες επιπτώσεις. Πώς θα διασφαλίσουμε τη βοήθεια που παρέχουμε πάει στους σωστούς ανθρώπους. Εγώ για χρόνια ασχολήθηκα με τα θέματα αυτά ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές πολέμου, στο Σαράγεβο και αλλού. Είναι τεράστια δυσκολία στο να προσπαθήσουμε να πετύχουμε να πάει στους σωστούς ανθρώπους η βοήθεια. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι μηχανισμοί, αλλά η πραγματικότητα που ισχύει επί τόπου είναι αρκετά περίπλοκη και δεν υπάρχει απόλυτα βέβαιος τρόπος να βεβαιωθούμε ότι η βοήθεια που παρέχουμε θα φτάσει στους σωστούς ανθρώπους. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό εκ των προτέρων, θα οδηγήσει σε αδράνεια. Και νομίζω κανείς δεν θέλει αδράνεια εδώ από τους παρόντες. Αν υπάρξει λοιπόν αν υπάρχουν αποδείξεις ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά βοήθεια, να τη δούμε. Να ενημερωθούμε και να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα βοήθειας. Επίσης, να συγχαρώ τον προλύσαντα, επειδή ήταν πολύ ξεκάθαρος για το γεγονός ότι δεν υπάρχει στρατιωτική νίκη στη Συρία. Υπάρχουν στρατιωτικά μέσα προς μια πολιτική λύση. Αυτό πρέπει να το παραδεχτεί κανείς και να αναγνωρίσει ότι το Ισλαμικό κράτος και η κατοχή εδαφών από αυτό είναι μια παγκόσμια απειλή που δεν πρέπει να επιτρέψουμε. Και αυτό βεβαίω επιφέρει μια στρατιωτική πτυχή. Αλλά δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σειρά της Συρίας. Και αυτό με οδηγεί στο αρχικό σημείο για τις διπλωματικές προσπάθειες και την χρήση κάθε πιθανής οδού ώστε να χρησιμοποιήσουμε τις υπάρχουσες διπλωματικές οδούς αλλά και τη βοήθεια και το capacity building που είχαμε μέχρι τώρα σε συνεργασία με τις διάφορες ομάδες που δρούν τοπικά. Να αναφερθώ και σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την διάσταση του CSDP. Εγώ δεν πιστεύω προσωπικά, γκλάδο και εκφράζομαι προσωπικά ότι υπάρχει λόγος για αποστολή σε SDP όσον αφορά τη Συρία. Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι έχει δυνατότητα η Ένωση μέσω του CSDP να κάνει κάτι. Αυτό είναι διαφορετικό πιστεύω, αναφέρθηκε, αλλά είναι και σημαντικό αυτό γιατί αν θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας την ευρωπαϊκή ασφάλεια τότε θα πρέπει εμείς πραγματικά να δράσουμε διπλωματικά και θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η Ευρώπη συλλογικά έχει δυνατότητα να αμυνθεί και πάλι το ένα δεν αποκλείει το άλλο δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ένα δίλημα είτε ανθρωπιστική βοήθεια και διπλωματική είτε στρατιωτική λύση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ένας ε, πάροχος ασφάλειας, θα πρέπει να έχει τα δικά της μέσα για να προσπιστεί την ασφαλεία της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω εργάζεται σε ένα σχέδιο δράσης άμυνας και ασφάλειας και αυτό έχει σημασία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση CSDP για κάθε πρόβλημα. Το ένα δεν αποκλεί το άλλο, το ξαναλέω, αλλά θα ήθελα να παραθέσω σε αυτά που είπε ο δηλαδή ότι έχουμε μια τεράστια περιπλοκότητα εδώ σε αυτά τα ζητήματα και να, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι έδειξε ηγετικά χαρακτηριστικά στο θέμα αυτό τις μέση Ανατολής, ε, στο θέμα της ε, συμφωνίας για τα πυρηνικά για το Ιράν, με το Ιράν που είχε τεράστια σημασία και αυτό αφορά μια χώρα που έχει τεράστιες πυρηνικές ε, δυνατότητες και τώρα έχουμε μια συμφωνία με τη διεθνή κοινότητα και η χώρα αυτή έχει απορρίψει επιθετική, οποιαδήποτε επιθετική στάση με τη χρήση πυρηνικών και εδώ σε αυτό το ζήτημα είχε κέριο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εικόνα λοιπόν είναι αρκετά περίπλοκη η γενική και εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει εμείς να είμαστε περήφανοι και να διαφημιζόμαστε παντού και πάντα πρέπει να παραδεχτούμε ότι εμείς ε, παρέχουμε βοήθεια για την ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια, ε, στήριξη η οποία είναι κρίσιμη σημασία και η συνολική δέσμευση της Ευρώπης και συμμετοχή σε διπλωματικό επίπεδο τώρα, αν ήταν υπαρκής, δεν ξέρω. Είναι δύσκολο βέβαια να πει κανείς ή να ισχυριστεί ότι είχαμε ομόνια η ομοφωνία στο θέμα της Συρίας. Όμως, όμως, η ευρωπαϊκή διάσταση μέσω CSDP ως απάντηση σε όλα τα προβλήματα νομίζω δεν καλύπτει και δεν αντιμετωπίσει σωστά το θέμα της Συρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Βεναμό, παρακαλώ έχετε το λόγο τώρα. Ευχαριστώ και πάλι. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια ερωτήματά σας. Να πέσω και στη Τζένι στο τέλος, γιατί νομίζω ότι πολλά από αυτά που είπατε αναφέρθηκαν, αναφέρονταν στην δικιά μου την παρέμβαση. Να συνοψίσω με τρεις τρόπους το τι μπορούμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε πραγματικά που πάει η βοήθεια. να κάνουμε και μια μελέτη αντικτύπου για τις επιπτώσεις των αντίπινων στην περίπτωση της Συρίας των κυρώσεων ξέρουμε όμως ότι το καθεστώς ε, Ασάντ χρησιμοποιεί αυτές τις κυρώσεις υπέρ του εις του πληθυσμού του Θα ήθελα εδώ να ξέρουμε περισσότερα πράγματα για τις επιπτώσεις επιτόπου της βοήθειας που προσφέρουμε και τις επιπτώσεις των κυρώσεων που έχουμε επίσης εφαρμόσει. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ήμουνα κι εγώ στα Βαλκάνια για μερικά χρόνια, πήγα και στο Αφγανιστάν και ξέρω ότι έχω χάσει λιγάκι την επαφή με το τι γίνεται επί τόπου. Κάποιος στην Κομισιόν μου είπε πριν από μερικούς μήνες ότι δεν είμαστε τυφλοί, δεν είναι τυφλή η Ευρώπη. Το 30% της Μέσης Ανατολής δεν γνωρίζουμε ε, τι κάνει, τι γίνεται με τα προγράμματα. Σε 30% των περιπτώσεων δηλαδή ότι χάνουμε την επαφή. Και τότε τι, να μην δράσουμε. Ε, μερικές φορές ναι, λέω, αλλά Άλλες φορές θα έλεγα καλύτερα να μην κάνουμε, να σταθούμε, να σκεφτούμε τις επιπτώσεις της βοηθειάς μας πρώτα. Το δεύτερο που θέλω να πω έχει να κάνει με την διαχείριση συνόρων. Άκουγα έναν στρατηγό Γάλλο να λέει ότι δεν έχει νόημα τώρα η ΙΤΑ της ΔΑΣ. Πρώτα πρέπει να έχει η Ευρώπη ένα καλό σύστημα διαχείρισης νόρων, γιατί αν τους καταστρέψουμε τώρα, θα έρθουν στην Ευρώπη πολύ γρήγορα. Και έχει δίκιο νομίζω. Κάποιοι θα σας πούν ότι η αντιμετώπιση μέσω της Τουρκίας βοηθάει την Ευρώπη να έχει ένα πιο ασφαλές σύστημα διαχείρισης νόρων. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η διαπραγμάτευση με την Τουρκία δεν μας οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση. Άλλοι όμως θα σας πούν ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Και το τρίτο που θέλω να πω, ναι, να δώσουμε περισσότερο περιθώριο σε άλλα μέσα. Λέτε ότι η ΚΠΑ δεν είναι ό,τι καλύτερο για να αντιμετωπιστεί η κρίση στη Συρία. Η ήμουν στη Γιούλεξ στο Κωσυφοπαίδιο για μερικά χρόνια και ποτέ δεν φαντάστηκα ότι μια αποστολή κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα θα βοηθούσε τώρα στη Μέση Ανατολή. Ακόμα και αν υπήρχε περιθώριο για την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα, θα σας πούνε όλοι ότι λειτουργεί με τέτοιους ρυθμούς δεν χρηματοδοτείται κιόλα με ένα σαφέ χρηματοδοτικό σύστημα που τελικά καμία χώρα δεν σκέφτεται να χρησιμοποιήσει αυτή την κοινή πολιτική, ακόμα κι αν ήταν εφικτό κάποτε. Αυτό δείχνει το που ακριβώς βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι δυνατότητες έχει να ανταποκριθεί. Το ίδιο μπορείτε να πείτε και για άλλες περιπτώσεις. Η συζήτηση για την κατάρτιση και τον εξοπλισμό επίσης χρειάζεται χρόνο για να αποφέρει καρπούς. Επί το που ξέρω ότι το συζητάτε αυτό στο Κοινοβούλιο τώρα. Πρέπει να επιταχυνθούν όμως οι συζητήσεις αυτές. Λοιπόν, συνοψίζοντας, λέω ότι ναι, για την βοήθεια που δίνουμε, σημείωσε αυτό που λέτε, διαχείριση συνόρων είπα, ε, περισσότερα κονδύλια για ε, το στρατιωτικό σκέλος, αλλά τα λέω όλα αυτά γνωρίζοντας πολύ καλά τι κάνουν οι άνθρωποι που δουλεύουν επί τόπου και προσφέρουν την ανθρωπιστική αυτή βοήθεια. Είναι φοβερή, είναι καταπληκτική. Αλλά δεν φτάνουν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο κύριος Μπροκ, είναι εδώ παρόν και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να ελευθερωθώ νωρίτερα είχα άλλες υποχρεώσεις. Άκουσα όμως μέρος της συζήτησης. Είναι μια κρόση αυτή που δημιούργησε αίσθηση και αυτό είναι πάντα θετικό. Είναι καλό σημάδι. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν υπό μια σύνθεση αρκετά κλασική. Ε, αφιβάλλουμε για αυτά που γνωρίζουμε, αφιβάλλουμε για τις ερμηνείες που ακούμε. Ε, βάλατε ζυζάνια εδώ. Δεν τα φέρατε εσείς όμως. Υπήρχαν. Γιατί ισχύουν όλα. Και βλέπετε ότι υπάρχει ένα τεράστια... Υπάρχει η άποψη που υπερισχύει ότι τίποτα δεν είναι πανάκι από μόνο του. Αυτή είναι η κλασική αντίθεση ανάμεσα στην Δύση και τη Ρωσία και στις Ηνωμένε Πολιτείες και στη Ρωσία. Υπάρχει το θέμα Ιράν και Σαουδικής Αραβίας και των ε, πολέμων διαντιπροσώπου. Έχουμε το θέμα της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου του Κουρδικού. Έχουμε την αντίθεση ανάμεσα στις ε, δυνάμεις της αντιπολίτευσης που είναι κατά του Ασάντε, της λεγόμενης καλής αντιπολίτευσης που προσπαθεί να πετύχει καλύτερες συνθήκες ε, σε συνέχεια της ε, Αραβικής Άνοιξης και απ' την άλλη έχουμε ομάδες όπως είναι η Αλκαΐδα και η Τζαπάτα Νούσρα. και έχουμε και την αντίθεση με το Ισλαμικό κράτος. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε εδώ πέρα διάφορες ε, αντιθέσεις οι οποίες ε, επικαλύπτονται και ε, εν μέρη φτάνουμε και σε πόλεμο. Και θα πρέπει να φροντίσουμε να τα, να τα βάλουμε όλα σε τάξη. Κατά τις επισκέψεις μου εκεί ε, τέθηκε επανειλημμένα το θέμα των μειονοτήτων. Ε, δεν ήμασταν σε θέση να προστατεύσουμε επαρκώς τις μειονότητες ε, που προστατεύονταν επαρκώς μόνο υπό το καθεστώς Ασάντ. Αυτό είναι γεγονός και ιδιαίτερα οι χριστιανοί. Θα πρέπει να εξεταστούν σε αυτό το πλαίσιο οι χριστιανικές εκκλησίες με πολλούς λογικούς ανθρώπους. Συνεργάστηκαν με τον ε, Ασάντ, ο οποίος ε, κατά τα άλλα ε, είναι άνθρωπος που έχει σκοτώσει πολλούς ανθρώπους επειδή αυτός τους προστάτευε. και υπόθηκε ότι πρέπει να υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη ώστε να στηρίξουμε τους μετριοπαθείς Σουνίτες αλλά οι μειονότητες αυτές δεν το πιστεύουν. Ε, αυτή είναι η θέση που ακούσαμε και στο Ιράκ και στη Μοσούλη και αλλού. Μας λένε πώς μπορούμε να επιστρέψουμε στις πόλεις μας ε, όταν θα επικρατήσει η ειρήνη. Ε, όταν ξαναδούμε τους ε, γειτόνους μας με τους οποίους ζούσαμε εν ειρήνη για κάποιο διάστημα αλλά από τη μία μέρα στην άλλη ε, ξαφνικά έγιναν διώκτες μας. έχει εξαφανιστεί λοιπόν αυτή η εμπιστοσύνη που υπήρχε. Και αλλού το έχουμε δει αυτό. Ε, τα παιδιά πηγαίνανε στο νηφιαγωγείο μαζί και από τη μία μέρα στην άλλη ξαφνικά ε, άρχισε ο κόσμος να πυροβολεί εναντίον των γνωστών του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, δεν μπορεί όμως να υπάρξει εάν δεν υπάρχει αξιόπιστη εγγύηση προστασίας απ' έξω. και μας ενδιαφέρει να ξέρουμε και τα σχετικά αριθμητικά στοιχεία. Το μήνυμα της Ρωσίας ε, ότι αποσύρεται ε, αφού έχει εξασφαλίσει τη θέση της εκεί ε, το μήνυμα αυτό ίσως είναι θετικό, αλλά ίσως ε, τώρα μπορέσουμε να αγωνιστούμε κατά του Ισλαμικού κράτους. Τι ακριβώς θέλω να πω. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εσωτερικές διαμάχες στη Συρία, την δυτική Συρία, ε, η πάυση πυρός ε, ανάμεσα στο καθεστώς ε, Ασάντ ε, και την αντιπολίτευση όλα αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε εάν έχουμε μία διαδικασία σε διάφορα στάδια. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην γίνεται πια πόλεμος και όλες οι δυνάμεις, είτε είναι οι διεθνείς δυνάμεις είτε οι περιφερειακές, θα πρέπει να είναι σε θέση να καταπολεμήσουν το Ισλαμικό κράτος ε, χωρίς ε, να επηρεάζονται από τις άλλες αντιθέσεις που υπάρχουν εκεί. Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα που υπάρχει για μια ειρηνική λύση. Κανένας ε, δεν βρίσκει καλό το Ισλαμικό κράτος, ούτε οι Ρώσοι, λόγω των ε, ε, Ισλαμικών δημοκρατιών τους. Ούτε οι Ιρανοί, ούτε καν οι Σαουδικοί Άραβες δεν βρίσκουν καλό το Ισλαμικό κράτος. Και γι' αυτό υπάρχει ενδεχομένως η ευκαιρία να το πετύχουμε αυτό. Οι αδυναμίες της Ευρώπης. Στην αρχή ήμουνα κάπως αισιόδοξο. Πίστευα ότι ε, η κυρία Μογκερίνη είχε καλή δουλειά ε, και σε σχέση με το Ιράν. Ε, μετά ξεκίνησαν οι συνομιλίες της Βιέννης. Επίστεψα ότι θα μπορέσουμε να παίξουμε ανάλογο ρόλο εκεί. Βρέθηκα στα περιθώρια του, της διάσκεψης ασφάλειας στο Μόναχο. Είχαμε την πέμπτη συζητήσεις, είχαμε μετά την η πυρός ε, το Σάββατο ο Λαυρόφ ε, το ανακοίνωσε αυτό. Συζητήθηκε ακόμα και η συνεργασία ε, σε στρατιωτικά θέματα ανάμεσα στην Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά βλέπουμε ότι Μετά από ένα τηλεφώνημα ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ομπάμα ε, αποσύρθηκαν ε, τα ρωσικά στρατεύματα, αλλά εμείς δεν είχαμε τίποτα να πούμε εκεί. Η κυρία Μογκερίνη είπε ότι παίζουμε σημαντικό ρόλο, αλλά δεν παίζουμε ρόλο κατά την λήψη πολιτικών αποφάσεων. Όταν θέλει να δώσει κανείς ε, κάποιο κίνητρο, το κίνητρο θα λειτουργήσει μόνο ε, υπό την απειλή των κυρώσεων. Δεν έχουμε ε, στρατιωτικές ικανότητες και γι' αυτό δεν μας χρειάζονται. Για τους Αμερικανούς ε, και τους Ρώσους ε, βλέπουμε ότι έχουν πάρα πολλές ε, πληροφορίες και εμείς δεν υπήρξαμε παράγοντας, ούτε γίναμε παράγοντας καθότι η Γαλλία επικαλέστηκε το άρθρο 42-7 Δεν είχαμε συντονισμό. Οι Γερμανοί στείλανε μια αποστολή ε, επιτήρησης. Οι ε, Δανείοι στείλαν κάποια αεροπλάνα, αλλά δεν υπήρχε ούτε ε, ευρωπαϊκό αρχηγείο που να συντονίσει τις προσπάθειες. Τι, έγιναν, τι απέγιναν αυτές οι δραστηριότητες και γιατί δεν παίξαμε στρατηγικό ρόλο. Βοηθητικά στρατεύματα στείλαμε, δεν μπορέσαμε όμως να είμαστε μια πολιτική δύναμη που να συμμετέχει στο τραπέζι λήψης των αποφάσεων. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να παίξουμε σημαντικό ρόλο. Και είναι σημαντικές ε, για μας οι ανθρωπίνες ζωές, ε, οπότε ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε πρώτα να οικοδομήσουμε συνοριοφυλακή για να καταπολεμήσουμε το Ισλαμικό κράτος. Εάν τα ευρωπαϊκά κράτη συμφωνήσουν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες, τότε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τους ε, ε, τρομοκράτες και τους αλλοδαπούς πολεμιστές. Έχουμε τη Europol, μόνο πέντε κράτη όμως δίνουν όλες τις πληροφορίες που έχουν στην Europol για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η χώρα μου δεν ανήκει σε αυτές. Εφόσον λοιπόν ε, τα ευρωπαϊκά κράτη δεν μπορούν ε, ούτε να συμφωνήσουν ε, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, δεν πρόκειται να έχουν αξιοπιστία οι δράσεις μας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε και να στηρίξουμε αυτήν την γραμμή Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών και να δούμε τι δυνατότητες πρέπει να οικοδομήσουμε εμείς. Thank you, uh, Ευχαριστούμε, Πρόεδρο. Κύριο Φρανζουλίτς, έχει ζητήσει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα που προφανώς είναι πολύ δύσκολο να το συζητήσει κανείς σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Μιλώντας για τη Συρία, μπορούμε να πάμε πίσω πολλά χρόνια πριν όταν οι σπόροι των μελλοντικών συγκρούσεων φυτεύονταν στο χώμα εκεί. Όταν το Ιράκ φτιάχτηκε μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μασούλ μέχρι το 26 ανήκε στην Τουρκία, όταν ο Κεμάλ Αρτατούρκ την έδωσε στο νέο σχηματιθέν Ιράκ και άλλες περιοχές που τότε ανήκαν στη Συρία τώρα βρίσκονται σε άλλες χώρες. Σκεφτείτε λοιπόν τις μειονότητες και άλλων χωρών των περιοχών. Οι σπόροι των συγκρούσεων αυτών είναι πάρα πολύ παλιοί. Μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ευρώπη δεν ήταν τόσο αποφασιστική και αποφασισμένη να βάλει τάξη, κυρίως στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική που ήταν οι κύριες πύλες προς την Ευρώπη. Κυρίε και κύριοι, η περιοχή το Κύπρος και οι μας, Συρία, Ιράκ, κάποιος καφές χύθηκε, φέρνει τύχη, λέει ο κύριος Φραντζουλίτσα. Η κατάσταση λοιπόν έγινε σαν τον πύργο της Βαβέλ, που είναι στη Μεσοποταμία, στη Μεσοποταμία και το Ιράκ. Ναι, Βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες τάσεις σήμερα για να ηρεμήσει η κατάσταση. προκειμένου να στηριχτούν οι συνομιλίες μεταξύ των διαφόρων πλευρών στη Συρία. Το ίδιο όμως πρέπει να γίνει και στο Ιράκ. Γιατί βλέπετε αυτά που έγιναν με τη νέα κυβέρνηση δεν πρόσεξαν αρκετά τα δικαιώματα των Σουνιτών του Ιράκ. Ήταν εσύτες λέγονται μειονότητα, αλλά είναι 10 και 11 εκατομμύρια στο Ιράκ. Θα έπρεπε λοιπόν να ληφθούν και αυτοί υπόψη. Όλες λοιπόν αυτές οι χώρες της Μέσης Ανατολής θα έπρεπε να συμμετάσχουν σε μια διεθνή διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή με τη συμμετοχή, και αυτό πρέπει να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή λοιπόν όλων των χωρών της περιοχής και τη συμμετοχή των μεγάλων δυνάμεων. Μια διεθνής διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή. Αυτή η διάσκεψη θα έπρεπε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, να φτιάξει τις σχέσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής, να διασφαλίσει πολιτικές και οικονομικές συναλλαγές, την πολιτική κατάσταση, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των χριστιανών για παράδειγμα στο Ιράκ και τη Συρία που εξαφανίζονται σιγά σιγά και υπάρχουν και σε κι άλλοι. Χρειάζεται και ένα σύστημα εγγύσεων μεταξύ των χωρών στη Μέση Ανατολή. Με τη συμμετοχή όλων αυτών των χωρών και το Ιράν και την Τουρκία και τη Συρία, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, Λίβανο, Ιορδανία κλπ. κλπ. Είναι αναγκαίο κάτι τέτοιο. Αλλιώς υπάρχουν τόσοι πολλοί σπόροι ακόμα για πόλεμο και διαφωνίες που θα χρησιμοποιηθούν είτε από τις περιφερειακές δυνάμεις είτε από τις παγκόσμιες. Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι, είδαμε ότι η Αραβική Άνοιξη τελικά δεν ήταν Άνοιξη. Δεν ξέρω αν είναι φθινόπορο, μάλλον χειμώνας έγιναν. Δεν είδαμε εξελίξεις υπέρ της δημοκρατίας, κράτους δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα πολιτών, μειονοτήτων κλπ. Όλα αυτά δεν έγιναν και θα έπρεπε. Η Τινησία ίσως είναι η καλύτερη περίπτωση, αλλά και ακόμα στην περίπτωση της Τινησίας υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά να γίνουν. Και υπάρχει μια ένα το που λέει ότι όποιος πάει στη Συρία βλέπει ότι η Συρία επηρεάζει τα πράγματα παγκοσμίως, όχι μόνο στην περιοχή. Πρόεδρος, Τώρα, παρακαλώ, αν θέλετε να απαντήσετε πρώτα εσείς, κυρία. Ευχαριστώ. Ναι, για τις τελευταίες παρατηρήσεις. Λοιπόν, πρώτον θέλω να υπογραμμίσω ότι τέτοιες συζητήσεις σαν και αυτή είναι πολύ σημαντικές και είναι σημαντικό να ακούμε τις απόψεις που ακούσαμε, ακόμα και εκείνες που είναι κατά των όσων λέμε, γιατί όλες οι φωνές βοηθούν να πάμε μπροστά. Δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις έτσι κι αλλιώς, έτοιμες λύσεις. Πολύ ωραία θα ήταν. Αν υπήρχαν θα τις είχαμε ήδη βρει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αντιμετωπίζουμε, είμαστε αντιμέτωποι με μια πάρα πολύ βαθιά κρίση στη Μέση Ανατολή. Είναι κρίση της μορφής διακυβέρνησης, της εκπροσώπησης του κόσμου και η κρίση αυτή δεν πρόκειται να επιληθεί γρήγορα, δυστυχώς. Ελπίζω, ειλικρινά, η κατάπαυση πυρώσεως στη Συρία να οδηγήσει σε έναν διακανονισμό στην ειρήνη, παρόλο που είναι δύσκολο, και ό,τι και αν γίνει τελικά στο πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον κόσμο στη Μέση Ανατολή για να βοηθήσουμε και να καταλάβουμε τι μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Να δουλέψουμε πάνω στη διακυβέρνηση και να βοηθήσουμε τον κόσμο να ξαναβρει μια αξιοπρεπή ζωή, να μπορεί αξιοπρεπώς να κερδίσει. Αυτό πρέπει να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε για να υπαγορεύσουμε σε κανέναν τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσει εφ' εξής. Δεν είναι αυτό που έχουμε υπόψη μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ με αυτό. Θα ήθελα να προσθέσω ότι δεδομένων των όσων είπε και ο κύριος Μπροκ πρώτον δεν μιλάω για αμυντική στρατηγική αλλά σαν προτεραιότητα Θέλω να καθιστάσω τους πολίτες για το ότι έχουμε μια προστατευμένη περιοχή Σέγγεν. Αυτό είναι που μας βοηθάει να είμαστε δυνατοί παίκτες στην περιοχή. Το ότι δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε τα σύνορά μας είναι κάτι βέβαια που μας καθιστά πιο αδύναμους στα μάτια των υπολείπων. πριν προβάλλετε κάτι στο μέλλον, πρέπει μέσα σας να είναι αρκετά δυνατό. Και αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Εσείς, για παράδειγμα, αναφερθήκατε σε μια μαγική λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση με την σημερινή εξουσία. Όλοι οι παράγοντες επιτόπου νομίζουν ότι με τη βία θα λυθεί το πρόβλημα, στρατιωτικά δηλαδή. Συνεπώς, πρέπει να περιμένουμε περισσότερη καταστροφή πριν μια τέτοια διάσκεψη λάβει χώρα με συμμετοχή των διαφόρων παραγόντων. Συνεπώς, νομίζω ότι καταρχήν είναι τα σύνορα και στη συνέχεια πρέπει να ανακτήσουμε εμπιστοσύνη στη στρατιωτική μας δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες ε, διότι μια τέτοια συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Η κατάσταση είναι τόσο πολύπλοκη και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να τη συζητούμε ε, συνέχεια εκ νέου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Έλμαρ Πρόκ που κανόνισε να παρευρεθούν και οι εμπειρογνώμονες. Μπορούσαμε λοιπόν να ακούσουμε διάφορες απόψεις. Τονίζουμε το θέμα των μειονοτήτων και ιδιαίτερα των χριστιανών. Αλλά φοβάμαι ότι ο Πασάρα Λασάντ και η κυβέρνηση της Συρίας εδώ και πολύ καιρό αποφάσισε να μην βασίζεται στις μειονότητες, όπως συνήθιζε, αλλά να επικεντρωθεί στην ε, μεγάλη ε, ε, αντίθεση ανάμεσα στους Σιήτες και τους Σουνίτες. Δεν είμαι απόλυτα πεπισμένη γι' αυτό, αλλά κάπως έτσι φαίνονται τα πράγματα. Κύριε Μπρόκ, συμφωνώ και με τη θέση σας. σχετικά με την ε, αλληλουχία των γεγονότων. Δεν υπάρχει κενό στην πολιτική. Είδαμε τι έγινε και στην ε, Σρεμπρενίτσα. Η διεθνής κοινότητα συχνά φοβάται να μην επέμβει. Τι θα γίνει αν δεν επέμβει σε, σε τέτοιο ε, περιστατικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους ε, συμμετέχοντες στη συζήτηση και ιδιαίτερα τους εμπειρογνώμονές μας. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ καθίστε. Please be seated. We have... Καθίστε παρακαλώ, έχουμε ακόμα δύο σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξή μας. Το επόμενο θέμα. διακόπτει πρόεδρος. Poproszę Θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε ησυχία, παρακαλώ. Ησυχία και καθίστε. Ξεκινάμε το επόμενο σημείο της ημερησίας μας. Δεύτερη συζήτηση για την έκθεση πρωτοβουλία, σχετικά με τι διαστημικέ δυνατότητε για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Η συγγητής, ο κύριος Μπόγκταν Ζντρογεύσκη, εκ μέρου τη Ήτρε, η συγγητής είναι ο κύριος Μαρινέσκου, Σκιώδη. έχουμε από όλε πολιτικές ομάδες, και η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι, ήταν 23 Φλεβάρι τον περασμένο μήνα. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή, στον κύριο Στρογεύσκη. Παρακαλώ κύριε Στρογεύσκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και έχουμε δύο εκθέσεις ακόμα. Οπότε να είμαι σύντομος να σας ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή έλαβα γύρω στι 200 τροπολογίες τροπολογίες οι οποίες διευρύνουν το θέμα και πάνε στη σωστή κατεύθυνση και αυτό είναι κατανοητό γιατί αν δούμε τα δορυφορικά συστήματα που κοστίζουν πολλά δις ευρώ τότε θα θέλαμε αυτό να είναι όσο πιο αποτελεσματικό γίνεται και να αντιμετωπίσουμε διάφορε προκλήσεις, όχι μόνο οικονομικές και ασφάλειες, αλλά και άλλες προκλήσεις. Και πρέπει να ομολογήσω ότι οι περισσότερες από τις τροπολογίες σας απευθύθηκαν σε μένα προσωπικά ακριβώς για να βελτιώσω την λειτουργία όλων αυτών των στοιχείων. Έλαβα λοιπόν και κάποιες παρατηρήσεις από τον κύριο Μαρινέσκου σε σχέση με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων όσον αφορά τα δορυφορικά συστήματα ώστε να περιληφθούν θέματα που αφορούν την ανάπτυξη. Έκανα δεκτές όλες αυτές τις τροπολογίες, ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχουμε περιλάβει μια σημαντική οικονομική πτυχή στο σχέδιο της νομοδότησης, της έκθεσης αυτής μάλλον. Και με τη δουλειά που κάναμε μέχρι τώρα, μπορέσαμε να συντάξουμε 25 συμβαστικές προτάσεις που περιλαμβάνουν τις μεσές τροπολογίες που έλαβα. Οπότε η δουλειά μας θα είναι πιο εύκολη. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτούς από εσάς που κατέθεσαν μεγάλο αριθμό τροπολογιών, Λογκζόν, Γκάλερ, Κοσουλίτσα. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά και να σας πω επίσης ότι χθες δουλέψαμε πάνω σε κάποιες από αυτές τις ε, διατάξεις και το περιεχόμενο της έκθεσης και έχουμε πρόοδο. Ο κ. και επίσης ε, χθες στην συνεδρίαση με βοήθησε για να προετοιμάσω το κείμενο σε διάφορα τμήματά του. Συμφωνούμε όλοι το ότι τα ευρωπαϊκά συστήματα, Γαλλίο κτλ. είναι πάρα πολύ σημαντικά Οπότε θα πρέπει να ασφαλιστεί η χρηματοδότησή του. Τώρα βρισκόμαστε βεβαίω στην ε, φάση συγκεκριμενοποίηση τη δημιουργία αυτού του και ολοκλήρωση αυτού του δορυφορικού συστήματο, το οποίο όμω απαιτεί ισχυρέ εγγυήσει ώστε να χρησιμοποιηθεί δηλαδή με το σωστό τρόπο το δορυφορικό αυτό σύστημα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποιοι δορυφόροι έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωή κάποιοι όπως το Γαλιλαίο έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωή, άλλοι όπως ο Κοπέρνικος έχουν πιο σύντομη διάρκεια ζωή. Οπότε χρειαζόμαστε νέους δορυφόρους σε τροχιά. Θα πρέπει να πέρασουμε λοιπόν σε μια νέα φάση μετά το Κοπέρνικο και το Γαλιλαίο. Να σας ευχαριστήσω που περιλάβατε αυτό το σύστημα πάντω το θέμα εδώ, γιατί αυτό το σύστημα έχει τεράστια σημασία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και θεωρώ προσωπικά ότι για αυτό το θέμα υπάρχει κατανόηση από τους περισσότερους ε, ευρωβουλευτές και τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, αυτό να σας πω. Ευχαριστώ, λέει και Πρόεδρος. Έφτασε και ο κ. Μαρινέσκου. Μήπως θα θέλατε να λάβετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε την θέση σας. Παρακαλώ, ευχαριστώ Πρόεδρο Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Για την έκθεση δεν έχω παρατηρήσεις. Να να προσθέσω μόνο κάτι για το CSTP πρέπει να ενισχυθεί και το διάστημα θα πρέπει να περιληφθεί στη στρατηγική για το CSTP. Για την νομοδότηση τώρα θεωρώ ότι έχουμε περιλάβει τη θέση της βιομηχανίας της δορυφορικής και θέλουμε το διάστημα ξαναλέω να περιληφθεί εδώ Έχουμε κάποιες θέσεις, έχουμε το εργαλείο το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί και για θέματα ασφαλείας και να κάνουμε τα απαραίτητα ώστε να είναι χρήσιμο το εργαλείο σύστημα και για ασφάλεια και για άμυνα. Έχουμε το Κοπέρνικους αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη ευκρίνεια και για την κυβερνοασφάλεια χρειαζόμαστε απαραίτητα για να προστατευτούν αυτά τα συστήματα. Προτείνουμε κάποιες αναλλακτικέ λύσεις με ένα νέο σύστημα για την Ευρώπη, ένα άλλο σύστημα δηλαδή το οποίο θα χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες δυνατότητες μαζί με κάποιες νέες ίσως και βεβαίως χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο θα αποτελείται από δυνατότητε οι οποίες υπάρχουν στο εμπόριο. Υπό μια διακυβέρνηση βέβαια για την οποία και για αυτήν κάνουμε κάποιε προτάσεις. Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε ένα SSD, ένα σύστημα δηλαδή το οποίο θα προστατεύει όλο, όλα τα συστήματα που είναι σε τροχιά στο διάστημα και τα διάφορα απορρίμματα που υπάρχουν γύρω από τους δορυφόρους. Και αυτό λοιπόν το σύστημα θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό ευρωπαϊκή διακυβέρνηση για να προστατεύει αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε για το μέλλον. Ζητάμε λοιπόν χρήματα για έρευνα και κοινοδομία βεβαίως και την ανάπτυξη του Γαλλίου και του Κοπέρνικου και για τα επόμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλοι και η Πρόεδρος. Κύριος το Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχά επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον εισηγητή. Είναι εξαιρετική αυτή η έκθεση. Ταυτόχρονα θα ήθελα να επιδιώξω την συμπερίληψη των τροπολογιών μας ε, στον συμβιβασμό Μάλλον συμφωνήθηκε χθε ο συμβιβασμό και ελπίζω ότι ε, αυτό θα οδηγήσει σε ευρία υποστήριξη τη έκθεση αυτή ε, στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να επαναλάβω την δέσμευσή μας να αποφύγουμε πλήρη στρατιωτικοποίηση ε, του τομέα και θα θέλαμε η πατή εκπρόσωπος να ασχοληθεί με το θέμα. Επιπλέον επικροτώ την αναδιατύπωση της παραγράφου 19. Ε, ε, συμφωνήσαμε να αναπτυχθεί το αναγκαίο χρηματοδοτικό πλαίσιο ε, να συμπεριλάβουμε δηλαδή αυτή τη διατύπωση, διότι έτσι πιστεύουμε ότι και οι εταιροί μας θα δεχτούν καλύτερα την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ε, για την ε, ανάπτυξη των ε, διαστημικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, όσον αφορά την στρατηγική αυτονομία, παίζει θεμελιώδη ρόλο απέναντι στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη ως προς την ασφάλεια. Θα πρέπει να έχουμε σαφή στρατηγική και θα πρέπει να φροντίσουμε να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις για να πετύχουμε τον στόχο μας. επενδύσεις στο σύστημα Γκαλιλαίου θα πρέπει να γίνουν ε, εάν θέλουμε να βρισκόμαστε σε ίδιο, στο ίδιο επίπεδο με άλλους διεθνείς παράγοντες ε, στο μέλλον όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, το ΝΑΤΟ και τη Ιαπωνία είναι πιο σημαντική από ποτέ για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το τεχνολογικό χάσμα που υπάρχει. Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη θα πρέπει επίσης ε, να είναι μεγάλη δύναμη. Είχαμε την ε, συζήτηση για τη Συρία, αλλά η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να συμμετέχει σε αποφάσεις εάν δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα εξωτερικά της σύνορα. Έχει μειωθεί πολύ ο ρόλος μας και αυτό θα συνεχίσει να ισχύει εάν δεν καταφέρουμε να οικοδομήσουμε μια πραγματική κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και δεν οικοδομήσουμε πραγματικές δυνατότητες άμυνες. Η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις απειλές και τις προκλήσεις του μέλλοντος η κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί στον τομέα της ε, κοινή ασφάλειας και άμυνας ε, και όπως γνωρίζετε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ε, βασίζονται κυρίως στο ΝΑΤΟ για την ασφάλειά τους, αλλά έχουμε δει ότι η παλαιά πολιτική του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μας έφεραν επιτυχία. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, καθώς ε, και τον εισηγητή που ήταν ανοιχτός απέναντι σε όλες τις απόψεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην έκθεσή σας αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κρασνατεύσκη, παρακαλώ. Σκιώδης εισηγητής του ECR. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ καλή η έκθεση αυτή. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Στρογεύσκη ε, για την συνεργασία σας ε, και που ε, υιοθετήσατε κάποιες από τις τροπολογίες μας. θα ήθελα να τονίσω τις δύο ιδέες που θέλετε να συμπεριλάβετε που είναι και οι πιο σημαντικές για μας και που αναφέρονται στις τροπολογίες μας. Καταρχάς, η ιδέα της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ρωσία στον ευαίσθητο αυτόν τομέα, στο Κοπέρνικους ε, και, ε, τα και τους δορυφόρους ε, που εκτοξεύονται με πύραυλους Σογιούς. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τη σχετική διατύπωση. Η κυρία Γκόμες ε, είχε μια έκθεση της 12ης Μαΐου του 2015. 15 όπου αναφερόταν ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τον αντίκτυπο διαφόρων προγραμμάτων στην αυτονομία και ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η συνεργασία με τη Ρωσία σε ε, τομείς όπως είναι η εκτόξευση πυράβλων Σογιούς ε, είναι ένα από αυτά. Ίσως θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Η δεύτερη μου παρατήρηση που νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σχετίζεται με μια από τις τροπολογίες μας όσον αφορά τη συγκέντρωση της, βιομηχανίας, ε, της διεθνικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Ε, το 70 και 90% αντίστοιχα των θέσεων απασχόλησης ε, συγκεντρώνονται σε ελάχιστες χώρες στον τομέα ε, του διαστήματος ε, και πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο να αναφέρεται αυτό στην έκθεση. Να συμμετέχουν δηλαδή περισσότερες χώρες και περισσότερες επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της υπερβολικής συγκέντρωσης. Νομίζω ότι πολλές χώρες μπορούν να επωφεληθούν Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να τους περιλάβουμε αυτό στην έκθεσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι άλλοι σκιώδεις εισηγητές δεν είναι παρόντες νομίζω. Έχω δίκιο, ναι πράγματι. Η γραμματεία μου το βεβαιώνει Προτού να ε, δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Βανόρτεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνο με τα περισσότερα από όσα είπε ο κύριος Κρασνοτεύσκη και είμαι ευγνώμων στον κύριο ε, που συμπεριέλαβε τις περισσότερες τροπολογίες μας ε, στο συμβαστικό κείμενο. Θα ήθελα να αναφερθώ στο, στη στρατηγική αυτονομία, κάτι που ακούμε συνέχεια. Δεν το καταλαβαίνω πολύ καλά Οι δημοκρατίες της Δύσης θα πρέπει να συνεργάζονται όταν υπάρχει στρατιωτική απειλή. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ιδιαίτερα όσοι μιλάνε για στρατηγική αυτονομία και από την άλλη θέλουν να εκτοξεύσουν ε, ε, τους, τους δορυφόρους μας με ε, ρωσικούς πυράβλους. Μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καθότι δεν βλέπω να είστε κανείς άλλο το λόγο, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Στρογεύσκη και στον κύριο Μαρινέσκου για να απαντήσουν. Σας ευχαριστώ και πάλι. Θα ήθελα να σας πω ότι βρίσκω ότι είναι Εξαιρετική η κατάσταση όσον αφορά τους δορυφόρους. Έχουμε την έγκριση από πολλές ομάδες που συνήθως έχουν διαφορετικές απόψεις. Έχουμε λάβει ε, προτάσεις από όλους αυτούς. Θα ήθελα να πω ότι η συμβολή του κυρίου Μαρινέσκου ήταν ιδιαίτερα ε, πολύτιμη. Και θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή. Η τεχνολογία των δορυφόρων θα πρέπει να ωφελήσει την Ευρώπη και την οικονομία μας. Ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε οικονομικά την Ευρώπη και νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται από όλους εδώ στην αίθουσα. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να συμπεριλάβω όλα τα στοιχεία που ανέφερε ο κύριος Κρασνοντέψκι και ε, θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Φανόρντεν και εγώ έχουμε επισημάνει συγκεκριμένους τομείς στην έκθεση για να πετύχουμε την ισορροπία ανάμεσα στα θέματα που αφορούν την άμυνα. Και η τελική μου παρατήρηση είναι ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα δύο διευθύνσει ε, που χειρίστηκαν το θέμα, αντιμετώπισαν το θέμα με ε, επαγγελματισμό. Φαίνεται να υπάρχει μια τάση αποκέντρωση, Μάλλον επιβραδύνεται η τάση συγκέντρωση. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Μαρινέσκου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να πω ότι στη γνωμοδότησή μας ε, μιλάμε για την ε, αυτονομία κατά την εκτόξευση. Ε, λέμε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να πετύχουμε αυτού του είδους την αυτονομία και αν θυμάμαι καλά Μόνο μία εκτόξευση θα γίνει με Σογιούς και τώρα το φθινόπωρο θα ξεκινήσουμε με ε, τους πυράβλους Αριάν και θα εκτοξεύσουμε τέσσερις πυράβλους. Έχει βελτιωθεί λοιπόν η κατάσταση στο συγκεκριμένο θέμα. Όσον αφορά την ε, σχετική βιομηχανία θέλουμε να παραμείνει στην Ευρώπη διότι είναι πολύ σημαντικός τομέας. Και βέβαια όλα εξαρτώνται από τη δυνατότητα κάθε κράτους μέλους να υποστηρίξει τέτοιες εργασίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φανζολίτσα. Ήθελε το λόγο. Ο εισηγητής ε, θα πρέπει να μπορεί να παρέμβει μετά για να απαντήσει. Ε. Ναι, Απλώς θέλω να τονίσω κάτι μετά από αυτά που είπε και ο κύριος Φανόρδεν. Ναι κύριε Φανόρδεν, εμείς βασίζουμε την ασφάλεια και την άμυνά μας στο ΝΑΤΟ. Συγχρόνως όμως λαμβάνουμε υπόψη μας ότι η προσφυγική κρίση χρησιμοποιείται πολιτικά από κάποιες χώρες. Ξέρετε, εκτός Ευρώπης για να προσπαθήσουν να αποσταθεροποιήσουν τον ευρωπαϊκό χώρο. Έχουμε μια κατάσταση στην Ευρώπη που δεν μπορεί η Ευρώπη να ελέγχει τα εξωτερικά της ε, σύνορα παραπάνω. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στον ΝΑΤΟ. Μερικές φορές τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν είναι τα ίδια με εκείνα του ΝΑΤΟ, οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αναπτύξουμε την ευρωπαϊκή ικανότητα για να ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους προκλήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε δεν θέλετε να... Για το διάστημα, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά χρειάζεται αυτονομία και διαστημικές ικανότητες, συμπληρωματικά όμως με τις δυνατότητες που έχει το ΝΑΤΟ. Πρόεδρος, καλώς. Κυρίες και κύριοι. Έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η δεύτερη εξέταση της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας για τις διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Σας υπενθυμίζω ότι η γνωμοδότηση της Ήτρε θα εγκριθεί στις 7 Απριλίου εκεί. Θα ψηφιστεί και στην ΑΦΕΤ θα ψηφίσουμε στις 17 στις 18 Απριλίου. Και στην Ολομέλεια θα πάει το θέμα τον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και αυτό το θέμα και έχουμε και άλλη μια έκθεση για σήμερα, που είναι επίσης έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. και επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης και συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και την Αφρικανική Ένωση. Είναι η δεύτερη εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Υπάρχουν οι σκιώδες οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Φανόρτεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τους και όδες εισηγητές και όλους τους συναδέρφους για τη συνεισφορά τους στην έκθεση αυτή. Όπως ξέρετε, θέλαμε η έκθεση αυτή να είναι ρεαλιστική. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνει στα πλαίσια, ανάλογα με τη συμβολή και των άλλων παραγόντων. Θέλω να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Πώς ε, να διαχειριστούμε περίπλοκες εταιρικέ σχέσεις, να αποφεύγεται η επικάλυψη των προσπαθειών, κατανομή έργου, να μην προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα κάνει όλα, αλλά να υπάρχει από αυτήν προσθεθέμενη αξία όπου μπορεί. Τονίζουμε επίσης και τη συμβολή των αφρικανικών χωρών γιατί όντω μπορούν να βοηθήσουν για την οικοδόμηση δυνατήτων, ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηγετικό ρόλο. Το APF, που είναι το Ταμείο εταιρική Αφρικανικής σχέση. Όσον αφορά την οικοδόμηση ικανοτήτων, είναι και αφρικανικές δυνάμεις που μπορούν να βοηθήσουν και έχουν βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη. Επίσης, η υποστήριξη όλων των πρεσβειών μας, των αντιπροσωπιών μας. Και αυτό προκειμένου να ενθαρρύνουμε τις αφρικανικές χώρες να αναλάβουν και εκείνες μέρος της ευθύνης. Τα κονδύλια που πηγαίνουν στην Αφρική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού να ελέγχονται επίσης από την Αφρικανική Ένωση. Είχαμε 120 τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Τις 67 τις έχω συμπεριλάβει στις συμβαστικές τροπολογίες. Θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω και τις κύριες ιδέες και τις προτάσεις και των υπόλοιπων συναδέρφων, αλλά φυσικά χωρίς να λιώνεται η ίδια φύση της έκθεσης. Γιατί η τροπολογία ε, από τις άλλες 53 τροπολογίες μπορώ πολλές να στηρίξω, 4, 5 και άλλες, αλλά είναι και μερικές με τις οποίες δυσκολεύομαι. Γιατί δεν έχουν σχέση με το θέμα της έκθεσης αυτής. Μερικές φορές εδώ οι συνάδελφοι προσπαθούν να προσθέσουν ε, πράγματα για να κάνουν έτσι προσωπικές σχέσεις. Δεν νομίζω όμως ότι είναι σωστό αυτό. Συνεπώς κύριε Πρόεδρε, αυτά εν συντομία είχα να πω εισαγωγικά και ελπίζω οι συνάδελφοι να στηρίξουν τις συστάσεις μου όταν φτάσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης είναι παρόν εδώ και ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Μάκιντας ονομάζομαι και ε, δουλεύω στο τμήμα Πανεπιστημιακών Σχέσεων. Ευχαριστούμε για το σχέδιο του κύριου Φανόρτεν όσον αφορά τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση Είναι ένα θέμα που σωστά συζητάει η Επιτροπή σας γιατί έχει να κάνει με την ανάπτυξη ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση είμαστε εταίροι υπέρ της σταθερότητας και της ειρήνης στην Αφρική και προωθούμε τις δραστηριότητες ειρήνης και ειρήνευσης όπου αυτό χρειάζεται. Η ειρήνη, ασφάλεια, συνεργαζόμαστε λοιπόν στα πλαίσια της εταιρικής μας σχέσης με την Αφρικανική Ένωση πάνω σε αυτά. Υπάρχει σημαντική οικονομική στήριξη στα πλαίσια της Αφρικανικής Διευκόλυνσης για την Ειρήνη που είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου. Τώρα υπογραμμίζεται πολύ η οικοδόμηση ικανοτήτων της ίδιας της Αφρικανικής Ένωσης με διάφορα συστήματα μεταξύ άλλων επικοινωνίες πληροφοριών κτλ. για να μπορούν να αντιμετωπίζουν από μόνοι τους οι Αφρικανοί κρίσεις. Η διευκόλυνση αυτή δίνει και θεσμική βοήθεια υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας. Για την οικοδόμηση ικανοτήτων στην Αφρική έχουμε πετύχει ήδη από τον Οκτώβριο που μας πέρασε με διάφορες ε, κοινέ δράσεις και τώρα τον Ιούνιο θα έχουμε διάσκεψη κορυφή όπου θα συζητηθεί ολόκληρο το θέμα των ικανοτήτων των δυνάμεων stand-by στην Αφρική. Προσπαθούμε λοιπόν να τους στηρίξουμε για την επίλυση των κρίσεων μέσω της προληπτικής ε, διπλωματίας και αποστολών. Οι αποστολές μας και οι δράσεις μας στην Αφρική βάσει της κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας συντονίζονται με την ΕΕ και την Αφρικανική Ένωση, ιδιαίτερα όταν ε, εκ παραλίλου συμμετέχουν και η Αφρικανική Ένωση όπως έγινε στη Σομαλία και στο Μαλί. Έχουμε επαφέ με την Αφρικανική Ένωση στα Ηνωμένα Έθνη και όχι μόνο στην έδρα αλλά και επί τόπου για να υπάρχει σωστή κατανομή εργατικού δυναμικού και για να αντιμετωπίζονται καταστάσεις συνειδητοποίησης και κατάλληλη ανάλυση. Και μια που μιλάμε εδώ πέρα για αυτά τα θέματα, θέλω να σας θυμίσω ότι υπογράψαμε διοικητικό διακανονισμό ανάμεσα Βακή Περισσία Εξωτερικής Δράσης και τις Συνεχτικές Δυνάμεις του ΟΗΕ με ανταλλαγή εγγράφων κτλ. Τα αναφέρω όλα αυτά γιατί το σχέδιο έκθεσης ε, μιλάει για την ολοκλήρωση αυτών των συμφωνιών ενώ έχουν αυτές ήδη υπογραφεί. Η δραστηριότητα αυτή είναι καρποφόρα όχι μόνο για περίπτωση κρίσεων, σε περίπτωση διαμεσολάβησης, αλλά και αφοπλισμού. Με την οικοδόμηση ικανοτήτων στην Αφρικανική Ένωση συζητάμε και με τα Ηνωμένα Έθνη. Πέρα από την Αφρική, στηρίζει η έκθεσή σας και τους στόχους της κενής δήλωσης για οικοδόμηση ικανοτήτων για ασφάλεια και άμυνα, προκειμένου οι εταίροι μας να μπορούν από μόνοι τους να αποφεύγουν ή να αντιμετωπίζουν κρίσεις, αλλά συγχρόνως στηρίζουμε και τις αρχές επιβολής του νόμου και τις στρατιωτικές αρχές στις χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τρογεύσκη. κυβέρνηση εκ μέρου του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταρχά να επιβεβαιώσω αυτό με το οποίο ξεκίνησε ο κύριος Πανόρτεν. Ρεαλιστική έκθεση και περιέχει κάποια στοιχεία επικριτικής προσέγγισης για κάποιες διαδικασίε στην Αφρική και λέει ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες όσον αφορά την αφρικανική πλευρά. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ αξιόλογο σχόλιο. Ώστε στην πλειοψηφία των σειράξεων να μπορέσουμε να μετατοπίσουμε έτσι την εστίασή μας προς αυτή την κατεύθυνση. Να τονίσω επίσης ότι καλωσορίζουμε την αποδοχή συμβαστικών προτάσεων και θα ήθελα αν απορρίψει κάποιες, να απορρίψει αυτές που δεν έχουν σχέση με την έκθεση, που δεν συνεισφέρουν δηλαδή σε σαφήνεια και σε σταθερότητα στο κείμενο. Και βεβαίω καταλαβαίνω αν ε, απορρίψει οποιαδήποτε άλλη η οποία δεν θα έχει σχέση με την έκθεση. Ευχαριστώ. Εισηγητή εκ μέρου των Σοσιαλιστών, παρακαλώ, και το λόγο. Ναι, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις για τις τροπολογίες και το κείμενο που δεχτήκαμε τον κύριο Πανόρθεν. Σχετικά με τις τροπολογίες που αφορούν την υπεραξία των Ευρωπαϊκή στην Αφρική, το θέμα των ευρωπαϊκών, συγγνώμη, των αφρικανικών στρατευμάτων και το αίτημα για νέα χρηματοδότηση για την αφρικανική δομή ειρήνης χρηματοδότηση που αφορά την αρχή ενίσχυση των Αφρικανών να ασφαλίσουν οι ίδιοι την ασφαλειά τους. Για τις συμβαστικέ προτάσεις, κάποιε παρατηρήσεις. Καταρχάς, για την γενικότερη ευρωπαϊκή πτυχή, η μορφή του κειμένου. Κάποιες αρκετέ ε, συμβαστικέ προτάσεις παρουσιάζουν, όπως η 16, μια αρνητική εικόνα της Ευρωπαϊκή παρέμβαση, άλλε ελαχιστοποιούν τη συμβολή αυτών των συλλογικών μα δράσεων η 1 και 2 και η 14. Ιδιαίτερα είμαι αντίθετος με οποιαδήποτε ιδέα που λέει ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να παρεμβληθεί στην ενίσχυση που θα μπορούσε να δει στην Αφρική. Μετά, για την γεωγραφική ισορροπία των δρασιών μας. Νομίζω ότι κάποιες από τις, αντιπροσω... από τις τροπολογίες μας έχουν ε, ενσωματωθεί στα εκτιμώντα όπως η 9. Παρ' όλα αυτά, η βασική ιδέα σύμφωνα με την οποία υπάρχει μια νέα τάξη ασφαλείας δεν εκπροσωπείται επαρκώς όπως η 93 τροπολογία που εγώ ίδιο συνέταξα και έστειλα. Είναι λοιπόν απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις κρίσεις με τρόπο ισορροπημένο για το σύνολο της Υπήρου. Και δεν είμαι υπέρ μιας εκ των προτέρων ε, διατύπωσης για χώρες προτεραιότητας σε εισαγωγικά όπως ε, προτείνει η συμβαστική πρόταση 5. Τρίτη πρόταση η σχέση μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης πολύ συχνά βρίσκεται σε δεύτερο πλάνο στις προτάσεις συμβασμού όπως η πρόταση 6 και 12. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να ενισχύσουμε τη διατύπωση εκεί επειδή δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα και ειρήνη χωρίς ανάπτυξη. Τέταρτη παρατήρηση. Όπως και άλλοι, για την 57 τροπολογία θεωρώ ότι θα πρέπει να επιδείξουμε κάποιο ρεαλισμό στις εξωτερικές μας δράσεις. Οι δράσεις μας θα πρέπει να καθοδηγούνται από τα συμφέροντά μας όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας. Νομίζω δεν χρειάζεται να δώσουμε την εντύπωση ότι οι αξίε μα είναι δευτερεύουσα σημασία, όπω ακριβώ προτείνει ο εισηγητή στα πλαίσια τη συμβαστική πρόταση 18. Η διατύπωση νομίζω είναι μάλλον ατυχή και θα ήθελα να αποσυρθεί. Πρόεδρε, αυτά από μένα και αγαπητοί συνάδελφοι, κάποιες παρατηρήσεις και δύο πρώτα λογάκια για αυτές τις συμβαστικές προτάσεις. Ελπίζω να διευκολύνω τον εισηγητή για τις μελλοντικέ φάσεις. Ευχαριστώ, πρόεδρο Πρόεδρος. Χαβιερ Βάστο, ο εισηγητής για την Άλτε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η σύνταξη το κ. Βανόρτε μου φαίνεται θαυμάσια επειδή είναι ρεαλιστική, επειδή νομίζω δίνει σωστέ ε, αναλογίες του συμβασμού μεταξύ των διαφορών ομάδων και νομίζω ότι καταβάλλει μια σημαντική προσπάθεια ώστε αντί να πάμε στους ασταθείς ωκεανούς της πολιτικής ορθότητας, να πάμε προς κάποιες πραγματικότητες τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Για την εφαρμογή της ειρήνης λοιπόν θα πρέπει να την σταθεροποιήσουμε και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε παρεμβάσεις και δράσεις για τη σταθεροποίηση της ειρήνης. Ιδιαίτερα εκεί όπου λείπει η ειρήνη και υπάρχουν τρομακτικές καταστάσεις. Παλαιότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια αφιλεγόμενη ουδετερότητα σταθερός και δεν πήγαινε πέρα της αστυνόμευσης, δηλαδή της διατήρησης της τάξης αφού αυτή υλοποιηθεί. Εδώ έχουμε κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα. Λέμε, ας πούμε, ότι δεν έχουμε μόνο τη μεταφυσική φιλοσοφική αξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά έχουμε μια ανυποχώρητη αξίωση σε σχέση με στρατιωτικές δομές οι οποίες αφού έχουν διαπράξει φρικαλαιότητες επιστρέφουν στις χώρες τους και δεν σημαίνει τίποτα. Εδώ πρέπει να έχουμε μια πρόθεση επαναφοράς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πέραν της πριτορικής. Ξέρουμε τι συμβαίνει σε διάφορες περιοχές όπου έχουμε διάφορες στατικές ομάδες που κάνουν διάφορες πράξεις και μετά επανέρχονται στις χώρες τους, γυρνάνε στις χώρες τους με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και δεν σημαίνει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Αυτό είναι γελίο νομίζω και έχει μεγάλη σημασία. Επίσης, καθορίζουμε μια καλύτερη διαλειτουργικότητα αυτών των αποστολών και όχι επικάλυψη. Υπάρχουν διάφορες δομές οι οποίες κάνουν την ίδια δουλειά πάλι στα πλαίσια ενό ε, ωκεανού διαλειτουργικότητα. Με εκθέσει οι οποίε μα ικανοποιούν θεωρητικά, αλλά δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα και να μιλήσω για τη δικιά μα επιχείρηση το Μαλί εκπαίδευση του στρατού του Μαλί εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν καταστροφικό γιατί μετά από δύο χρόνια εκπαίδευση δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε έναν λειτουργικό αξιόμαχο λόγο. Είναι... Ήταν απαράδεκτο αυτό. Δεν πετύχαμε τίποτα. Και έχει καλή την εντύπωση ότι όταν έχουμε να κάνουμε μια στρατιωτική επιχείρηση, αυτό γίνεται για να είναι αποτελεσματική αυτή η επιχείρηση. Όχι να μα ενημέρουν εδώ διάφοροι παρατρεχάμενοι για το τι συμβαίνει. Και όταν του ρωτάμε, αν εσεί έχετε σχηματίσει αυτό το λόγο, ο οποίο αντιμετωπίζει υποδεέστερε μονάδε είναι αποτελεσματικός και μάλλον είναι όχι. Τότε τι γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και να αξιολογούμε αυτά που συμβαίνουν. Μέχρι τώρα αυτό ήταν εξέχως απόν. Θεωρώ ότι θα συμφωνήσω με το επικριτικό πνεύμα του εισηγητή επειδή η κατάσταση απαιτεί ακριβώς σαφήνεια και σκληρότητα. Και να πω στον κύριο Βανόρτεν ότι δεν έχω συναντήσει συχνά άτομα που έχει τέτοια δυνατότητα αντίληψης και ανοίγματο των θέσεων του προς τους άλλους και με τεράστια δυνατότητα συνεργασίας. Για μένα η συνεργασία μαζί ήταν ε, απόλαυση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούζα. Σκεδούς εισηγητές εκ μέρους της Πρόεδρε, ευχαριστώ. θα σας στείλουμε μια έκθεση μειοψηφία πριν την ψηφορία. Γι' αυτό δεν έχουμε καταθέσει τροπολογίες, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Παλέρο, σκιώδης από τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω ότι έγινε πολύ καλή δουλειά μαζί με τον κύριο Φανόρδεν και νομίζω ότι είναι ισορροπημένο το κείμενο το οποίο επικεντρώνεται στα σημαντικά θέματα, όπως είπαν και άλλοι πριν. Εξέτασα τις συμβιβαστικές τροπολογίες που έλαβα σήμερα και χαίρομαι πολύ που έχουν υιοθετηθεί τόσες πολλές από τις προτάσεις μας. Δεν έχω εξετάσει όλες τις συμβαστικές τροπολογίες, δεν μπορώ να σας πω ακόμα πώς θα ψηφίσουμε, αλλά υποθέτω ότι θα έχουμε συνάντηση των σχεδόν εισηγητών ώστε να συζητήσουμε τις απόψεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων και να καταλήξουμε σε ένα καλοκείμενο. κείμενο. Ιδιαίτερα χαίρομαι για τη νέα παράγραφο 14α που αναφέρεται στην σεξουαλική εκμετάλλευση και abuse λέει ο ομιλητρία στα αγγλικά, κακοποίηση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το ότι έχει συμπεριληφθεί στην έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φανόρδεν και προσλέπω στη συνέχιση της καλή συνεργασία. Κύριε Φανόρδεν, θα θέλατε να απαντήσετε. Interventions. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εκτιμώ τις παρατηρήσεις ε, των συναδέρφων. Ε, είμαι ευγνώμων στον κύριο Νάρτ και την κυρία Βαλέρο για τις παρατηρήσεις τους. Καθώς ε, και στον ε, σκιωδή συγητή του ΕΛΚ. Πιο σημαντικό από όλα είναι να επικεντρωθούμε στην ουσία της ε, έκθεσης και ελπίζω ότι θα έχουμε μια συνάντηση σκιωδών εισηγητών για να συμφωνήσουμε. Νομίζω όμως ότι γενικά θα υποστήριξετε τις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Ε, υπάρχουν κάποια δύο μικρές δυσκολίες, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε λύση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι, ολοκληρώσαμε τη δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου έκθεσης του κυρίου Βανόρτεν. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η ψηφοφορία ε, προβλέπεται στις 18 Απριλίου στην ΑΦΕΤ και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Υπάρχει κάποιο θέμα υπό τα διάφορα. Εάν όχι, να σας θυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 20 και 21 Απριλίου. Σας ευχαριστώ.